Good morning, colleagues. Can I bring the meeting to order? Καλημέρα, συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε. next item on the agenda is the report. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη αναφορά για τα όσα έγιναν στην συνεδρία των συντονιστών χτες και ορισμός των ε, εισηγητών οι αποφάσει των συντονιστών έχουν ω εξή. Για τι νομοδοτήσει για τη δημιουργία του μηχανισμού για την Ευρωπαϊκή Γειτονία δεν ε, υπήρξε απόφαση από τους συντονιστέ. Για τις ε, ε, τεχνολογικές υπηρεσίες και τις μεταφορές, για τις δημόσιες προμήθειες, η απόφαση των συντονιστών ήταν να ενωθούν οι δυο αυτέ γνωμοδοτήσεις και να γίνει μία. Και θα την αναλάβει η ομάδα των Πρασίνων. Θα δώσει τον συντονιστή η ομάδα των Πρασίνων. Τώρα, για τα ε, ε, συμβάσει παραχώρησης, ε, η Γκουέ είπε ότι θέλει να αναλάβει την γνωμοδότηση τη σχετική για τις προτεραιότητες για το 2013 και τον, το τμήμα 3 του προπολογισμού. Η Κομισιόν θα θυμάται το κάνουμε αυτό ενημερωτικά μεταξύ των ε, ομάδων. Το 2013 θα πάει στο ALDE. Για τα έγγραφα που έχουμε λάβει τα ενημερωτικά, η ανακοίνωση της Κομισιόν και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό όραμα για τους ταξιδιώτες και τα δικαιώματα των επιβατών ε, στις μετακινήσεις τους, οι συντονιστές συμφώνησαν να ζητηθεί άδεια να γίνει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, μια γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας και αν αυτό γίνει αποδεκτό, τότε θα την αναλάβει το ΕΛΚ και θα δώσει τον εισηγητή. Για την ανακοίνωση της Κομισιόν για το μηχανισμό κινήτρων για την εφαρμογή του ΣΕΖΑ και, την, τον τεχνολογικό πυλώνα για τον ενιαίο ε, ενέργειο χώρο, είπαμε ότι θα υπάρξει συνεργασία για την υπάρχουσα γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η κυρία Φώστερ. Οπότε η κυρία Φώστερ θα το συμπεριλάβει και αυτό το κομμάτι στην γνωμοδότηση που έχει ήδη αναλάβει. Για, την, για τον ιστορικό κανονισμό της ε, Κομισιόν, για τα για, την ε, καλύτερη, ε, για το πιο καθαρό περιβάλλον περιμένουμε τι θα μας πει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Οπότε οι συντονιστές αποφάσισαν ότι θα περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα αποφασίσουν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Για τις, ε, για τις Επιτροπές Εργασίας για το 2010 οι συντονιστές είπαν να μην αναλυφθεί η δράση και για την ανακοίνωση της Κομισιόν για το πλαίσιο ισότητας για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Περιμένουμε την ΙΜΚΟ να λάβει απόφαση. Οπότε η απόφαση των συντονιστών είναι προς το παρόν να μην γίνει κάτι, να περιμένουμε τι θα πει η ΙΜΚΟ. Μετά, <coughs> τέσσερις εκθέσεις για το πακέτο για τις κρατικές επιχορηγήσεις ε, και το και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Η απόφαση ήταν να μην γίνει κάτι προς το παρόν. Μετά υπάρχει το πάνελ της ΤΟΑ. Οι συντονιστές ε, επιβεβαίωσαν την, ε, τον ορισμό του κυρίου Γκάνσιαν και της κυρίας Στικάου στο πάνελ της ΤΟΑ. Για τις μελέτες τώρα. Οι πολιτικές ομάδες θα στείλουν προτάσεις για μελέτες που θα γίνουν για την κατανομή του προπολογισμού του 2012. Η προθεσμία είναι Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι. Θα ληφθεί απόφαση μετά για το ποιε είναι αυτές οι μελέτες που θα προωθηθούν στην συνάντηση των συντονιστών στι 27 Φεβρουαρίου. Τώρα, για την επιτροπολογία. Οι συντονιστές εξέφρασαν τη λύπη τους για το ότι το σχέδιο εφαρμοστικών ε, και ε, ε, γραμμών για, το, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα για το 2012 το έλαβαν την προηγούμενη Πέμπτη. Και η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η ομάδα εργασίας μάλλον του Συμβουλίου, θα συναντήθηκε στις 20 του Γενάρη. Ε, αυτές οι πληροφορίες είπαν ότι πρέπει να δίδονται στο Κοινοβούλιο ε, σε, με ικανό χρόνο ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη και τα σχόλια που θα κάνει το Κοινοβούλιο στην τελική απόφαση. Η Κομισιόν λοιπόν θα ζητηθεί να παρουσιάσει τα μέτρα αυτά στην ε, συνάντηση των συντονιστών στις 6 Φεβρουαρίου και ζητήσαμε να εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον οι πληροφορίες αυτές θα μας αποστέλλονται με αρκετό χρονικό περιθώριο μπροστά μας ώστε να μπορούμε να τις μελετούμε. Στα διάφορα έχουμε την έκθεση follow-up για τις επιπτώσεις του κανονισμού του, του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Λάβαμε μία απόφαση το Νοέμβρη ότι το ΕΛΚ θα αναλάμβανε την γνωμοδότηση και θα πρότεινε έναν ε, εισηγητή για να γίνει μια ε, ίδιας πρωτοβουλίας ε, γνωμοδότηση από την Άγκρη. Ε, αλλά η Άγκρη δεν ξέρουμε αν θα κάνει ίδια, ε, δεν ξέραμε τότε αν θα έκανε ίδια πρωτοβουλία. Η Άγκρη είπε ότι θα αναλάβει την γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας, οπότε θα δώσει και τον εισηγητή για την ε, έκθεση αυτή. Τα μέλη θα γνωρίζουν ότι η προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πάντα είναι μεγάλο ζήτημα και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια σχετική γνωμοδότηση. Τώρα, οι αεροπορικέ μεταφορές, η αεροπλοεία στο, μπαίνει στο, κομμάτι, στο πακέτο για την ανταλλαγή εκπομπών. Ζητήθηκε από την Κομισιόν ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις. Και η Κομισιόν είπε ότι θα μας κάνει αυτή την ενημέρωση. Ε, η απόφαση αυτή δόθηκε και στους συντονιστές. Τώρα, το ψήφισμα για το GMES. Ε, Υπάρχει ένα ψήφισμα από την Ήτρε που δόθηκε στους συντονιστές ώστε να ληφθεί απόφαση αύριο για το κατά πόσο θα πρέπει ο πρόεδρος να στείλει μια υποστηρικτική επιστολή και το προτινόμενο κείμενο για την πειρατεία ε, θα κυκλοφορήσει ένα κείμενο σε όλες τις ομάδες με μια προθεσμία για τροπολογίες την 30 Ιανουαρίου το μεσημέρι ώστε να προχωρήσουμε μετά σε ό,τι αφορά την υποβολή προφορικής ερώτησης για το θέμα της πειρατείας. Αυτά από την συνεδρίαση των συντονιστών. Ερωτήματα ή σχόλια ή παρατηρήσεις υπάρχουν. Αν όχι, ευχαριστώ πολύ. Next item on the agenda. Επόμενο σημείο το μέλλον των υπηρεσιών αεροπλοείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μπράντουαρν έχει το λόγο που έχει αναλάβει και τη σχετική έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη ανταλλαγή που κάνουμε για το θέμα αυτό. Οπότε θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω γενικά για και να σας πω κάποια πράγματα για, τα... για τους πόρους που χρησιμοποίησα για να συντάξω αυτή την έκθεση. Τρία είναι τα, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι ύπαρξης αυτής της έκθεσης. Καταρχάς ο ορισμός, γιατί όπως το γνωρίζω εγώ, όπως το ξέρω, δεν υπάρχει α, ορισμός του τι είναι περιφερειακό αεροδρόμιο. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι ένα, ένα αεροδρόμιο που μπορεί να έχει κάτω από 5 ε, εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Κάποιοι λένε ότι είναι κάποιο ε, διαμετακόμισης αεροδρόμιο ή να έχει πολλές ε, συνδέσεις. Οπότε εγώ στην εκθεσή μου προσπάθησα καταρχάς να βρω έναν λογικό ορισμό για τους σκοπούς της καταγραφής των περιφερειακών αεροδρομίων και των υπηρεσιών βεβαίως που παρέχουν. Δεύτερον, να δούμε τις οικονομικές επιπτώσεις των περιφερειακών ε, αεροδρομίων και των υπηρεσιών τους. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι οι αεροπορικές υπηρεσίες ε, των που απορρέουν από τις περιφέρειες έχουν πολλές συνέπειες, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ύπαρξη θέσεων εργασίας, αλλά και σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάταξη, την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας που εξυπηρετούν. Και αυτό βεβαίως έχει και πολλαπλασιαστικές συνέπειες όσο αναπτύσσεται περισσότερο αυτό το αεροδρόμιο και οι υπηρεσίε του. Και το τρίτο σημείο ως γενική αρχή που προσπάθησα να μελετήσω ήταν ότι ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην έκθεση αυτή ειδικά σε τομείς που δεν ήταν ε, αποκλειστικοί για τα αεροδρόμια και τις υπηρεσίες τους, αλλά όπου η πολιτική στον τομέα αυτό της αεροπλοείας ε, έχει δυσανάλογες συνέπειες σε κάποιες περιπτώσεις σε αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκα όταν συνέτασα αυτή την έκθεση. Είδα και το θέμα λοιπόν, ε, είπα, σας είπα για τον ορισμό μάλλον. Ε, σύντομα θα ήθελα να πω και κάποια άλλα σημεία που προσπάθησα να τονίσω στην έκθεση. Τα οικονομικά, οικονομικές συνέπειες. Καταρχάς, τα περιφερειακά αεροδρόμια έχουν, είπαμε, αυτή την ε, πολλαπλασιαστική, τις πολλαπλασιαστικές συνέπειες ό,τι αφορά την οικονομία και κυρίως είναι εμπορικά αεροδρόμια, με εμπορικές δηλαδή δραστηριότητες. Εγώ λοιπόν προσπάθησα να δω ποιοι είναι οι τομείς της πολιτικής όπου υπάρχει είτε εθνική είτε ευρωπαϊκή νομοθεσία ή και εμπορική πολιτική η οποία να έχει αποβεί εις βάρος της ανάπτυξης των αεροδρομίων αυτών και των υπηρεσιών τους. Και αυτό ισχύει ειδικά σε ό,τι αφορά το πώ διαχειρίζονται τα αεροδρόμια τι ε, εμπορικέ δραστηριότητέ του. Και εγώ προσπάθησα να δω ποιοι είναι αυτοί οι τομεί που πρέπει να ε, επικεντρωθούμε και που, είναι τελικά, και που επηρεάζονται άδικα από την πολιτική που ε, επιβάλλεται για πολύ μεγαλύτερα αεροδρόμια των περιφερειακών. Επίσης, είδα αν υπάρχει συνδεσιμότητα μεταξύ των περιφερειακών αεροδρομίων και των υπηρεσιών τους και άλλων ειδών μεταφοράς. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε, Πρόεδρε, ότι σε κάποια κρατημέλη ε, κάποιες από τις εταιρείες, τις αεροπορικές, έχουν πολλαπλά εισιτήρια. Δηλαδή παίρνει κανείς ένα τρένο ειδικά στην Γερμανία και ουσιαστικά το τρένο αυτό έχει και έναν κωδικό αεροπορικό που το συνδέει με μια αεροπορική υπηρεσία. Αυτό πρέπει να το δούμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ε, δεν μιλούμε για ξεχωριστές, ε, ξεχωριστά είδη μεταφοράς. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε όλες αυτές τις ε, διαφορετικές μεθόδους είδη μεταφοράς. Οπότε εγώ θα ήθελα να δημιουργηθεί μια διαδικασία ώστε να μπορούμε να κλείνουμε ένα εισιτήριο από το αρχικό σημείο αναχώρησης μέχρι το τελικό σημείο άφηξης. Είτε είναι πλοίο, είτε είναι τρένο, είτε είναι σιδηρόδρομος, είτε είναι όλα αυτά μαζί. Οπότε είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Επίσης, Είδαμε και το πρόγραμμα TNT των διευρωπαϊκών δικτύων και θα θυμάστε ότι και πριν από χρόνια που κάναμε το πρόγραμμα την τελευταία φορά τα περιφερειακά αεροδρόμια συμπεριλαμβάνονταν από και οι υπηρεσίε του στο πρόγραμμα TNT και αυτό θα πρέπει να το δει η Κομισιόν ως τμήμα του δικτύου TNT. Από τότε βεβαίω λίγα έχουν γίνει από τότε που ενεκρίθη το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Δικτύων και θα ήθελα να επαναλάβω ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι σημείο κλειδί ε, στο όλο δίκτυο των ε, διευρωπαϊκών δικτύων που μελετούμε τώρα. Και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και ε, τις υπηρεσίες που παρέχουν αυτά τα ε, αεροδρόμια. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε και αν είναι ο τρόπο μεταφορά που επιλέγεται. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του πώ βλέπουμε το πρόγραμμα TEN-T. Τα σημαντικά περιφερειακά αεροδρόμια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ε, βασική στρατηγική. Επίση, είδα και κάποια θέματα διαφάνεια. Υπάρχουν και εκεί κάποια στοιχεία ειδικά σε ό,τι αφορά το, το κόστος για αυτά τα αεροδρόμια και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και που επηρεάζει τελικά αρνητικά την διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους επιβάτες που περνούν μέσα από κάποια ε, περιφερειακά αεροδρόμια για να πάνε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Επίσης, το θέμα των αποσκευών είναι σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι σε τα πιο μικρά αεροδρόμια χρησιμοποιούνται πιο μικρά αεροπλάνα. Οπότε δεν υπάρχουν κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ ώστε να μπορεί κάποιο να ξέρει ποια είναι η αποσκευή που επιτρέπεται να πάρει στο κάθε αεροσκάφο. αεροσκάφος. Οπότε και πάλι υπάρχει α, ασυνέπεια σε ό,τι αφορά τι επιπτώσει που έχει αυτό στι μικρέ αεροπορικέ εταιρείε. Αυτά, Πρόεδρε, έτσι γενικώ που τα στοιχεία που ανέφερα στην έκθεσή μου. Να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης και βεβαίως περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ, κύριε Μπράδο. Οι δύο βασικοί σκιώδεις συνεχές δεν έχουν έρθει ακόμα. Ο κύριος Ουτζίας κατευθείαν θα πάρει το λόγο. Ο κύριος Χέγγινς από το ΕΛΚ, καλύτερα, πρώτος, τον βλέπω, είναι εδώ. Ζητώ συγγνώμη. Θα μιλήσω εκ μέρους ενός άλλου συναδέλφου, ε, ο οποίος δεν είναι εδώ. Είναι θαυμάσια δουλειά που κάνει ο εισηγητής. Θέλω να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Καταρχάς, συμφωνώ με τα σχόλιά του ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ορισμό για τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρξει αυτός ο ορισμός. για το Recycle D. Σίγουρα οι λιανικές πωλήσει έχουν πάρα πολύ πέσει ε, από την εποχή που ε, μπήκαν αυτοί οι κανόνες. Καταρχάς, ε, οι καταναλωτές έχουν πληγεί. Ε, προσπαθούν να βάλουν όλες τις αποσκευές τους σε μία τις χειραποσκευές και τα λοιπά σε μία αποσκευή. Και επίσης πρέπει να πληρώσουν όλο και αυξημένες τιμές ε, για αυτά τα αεροδρόμια. Στην παράγραφο 21, οι κανόνες για το ποσό, το μέγεθος ε, της χειραποσκευής θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα για τις διαστάσεις των χειραποσκευών. Γιατί πολλοί ε, καταλαμβάνονται εξαπίνεις, Γιατί είναι είτε πολύ φαρδιές, είτε πολλές, πολύ μακριές, είτε πολύ στρογγυλές, είτε πολύ δεν ξέρω τι. Ε, και τελικά δηλαδή δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το ε, καλούπι με βάση το οποίο ε, μετράμε τις χειραποσκευές και επομένως δεν μπορούν να θεωρηθούν χειραποσκευές. Επίσης, για τους κοινού κανόνες σε ό,τι αφορά τα έξτρα κιλά και το πώς τα τιμολογούν οι εταιρείε. Ε, όμως, αφού η Ισπανική κυβέρνηση κατήρισε τον κανόνα του εις ε, μίας αποσκευής, μπορούν και άλλες ε, κυβέρνησεις να το κάνουν. Επίσης, οι δημόσιες υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχω όμω ε, επιφυλάξει την παράγραφο 13. Δεν ξέρω αν θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πληρώσουν για την επιπλέον ασφάλεια. Γιατί ούτω ή άλλως ε, πληρώνουν για τα τελωνία. Πληρώνουν για την αστυνομία. Για τον έλεγχο των διαβατήριων, Φερρυπίν. Και νομίζω ότι η ασφάλεια θα πρέπει να πληρωθεί από τα αεροδρόμια. Στην παράγραφο 20 Μ' αρέσει ε, ότι το γεγονός που λέτε κύριε εισηγητή, ότι θα πρέπει η τιμή που πληρώνει και που αναφέρεται στο εισιτήριο να είναι πιο διαφανής. Για τις πιστοτικές κάρτες και τις χρεωστικές κάρτες και το επιπλέον χρέος ε, στις, ε, στο 99% των πτήσεων, ακόμα και στην αγορά από ίντερνετ, χρησιμοποιούμε αυτές τις κάρτες. Ε, επομένως, θα πρέπει να επιτρέψουμε στις εταιρείες να, την υπερχρέωση. Αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί σε όλες τις μεθόδους πληρωμής. Δύο από τις ε, αεροπορικές μας εταιρείες, όπως η Ryanair, έχουν ένα είδος επιστοτικής κάρτας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις πτήσεις. Αλλά το πρόβλημα είναι είναι πολύ δύσκολο να τις έχουμε αυτές. Και επιπλέον ε, η υπερχρέωσή τους είναι πολύ μεγαλύτερη από τις... Επομένως, θέλω να βάλω μια τροπολογία στην έκθεση του κυρίου Μπράντμπορν. Ίσως το καλύτερο σημείο όμως είναι, ε, να το κάνω στην έκθεση για τα δικαιώματα των επιβατών. Κύριε Ισηγητά, ε, κοιτάξτε αυτά τα θέματα που είπα, ίσως για την απαγόρευση δηλαδή, των πιστοτικών καρτών. Τώρα, για το συνάδελφο που καλύπτω. Ε, ανησυχεί για τα νούμερα που υπάρχουν στην έκθεση. Και από πού ήρθαν αυτά τα νούμερα, λέει ο, μου λέει αυτός ο συνάδελφος, ανησυχεί. Για τον ορισμό των περιφερειακών αεροδρομίων, ε, εγώ όμως δεν συμφωνώ με αυτό που μου είπε ο συνάδελφος να πω, Τέλο πάντων, εγώ συμφωνώ ότι είναι καλός αυτός ο ορισμός των αεροδρομίων. Επίσης, ε, οι αεροπορικές εταιρείε λέει ο εισηγητής, ε, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα περιφερειακά αεροδρόμια. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Λέει ο κ. Σπίρκερ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ε, για τις επιπλέον χρεώσεις και για τα θέματα των, του συνδυασμένων μεταφορών σιδηροδρομικών και αεροπορικών. Ο κύριος Σασόλη δεν ε, χρειάζεται να σας πω εγώ ότι θα έρθει σύντομα οπότε θα, για να σας κάνει τα σχόλιά του, οπότε θα κάνω εγώ κάποια πολύ σύντομα σχόλια, τα οποία είναι αρκετά ουσιώδη βέβαια να ε, ευχαριστήσω τον κύριο Μπράτμπορν βεβαίως για την δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμή, Ήταν πραγματικά εξαιρετική. Ένα σημαντικό σημείο όμως είναι το εξή και το ανέφερε και ο συνάδελφος Higgins. Οι αεροπορικές εταιρείε προσπαθούν ε, αυτή τη στιγμή ε, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ε, ε, χειροποσκευές, να μειώσουν σημαντικά το μέγεθός τους, να εξοικονομήσουν χώρο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές εταιρείε που το κάνουν αυτό, αυτό έτσι ώστε στα, μέσα στα αεροπλάνα μπορούν να απολούν τα προϊόντα τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ενιαίες ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό, γιατί ήδη ανοίγονται αυθαίρετα διάφορες πόρτες που είναι πραγματικά τελείως αδιαφανείς για τους επιβάτες και δεν τους βοηθούν καθόλου, ούτε τους ωφελούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας και ειδικά της χρηματοδότησης για την ασφάλεια, δεν συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Higgins. Έχουμε μια έκθεση ήδη ψηφισμένη για την χρηματοδότηση των, της ασφάλειας των αεροδρομίων, όπου σαφώς αναφέρεται ότι τα μέτρα ασφαλείας ε, που ε, ξεπερνούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα μπορούν να χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη από, ε, από τους δικούς προπολογισμού. Ε, Βεβαίω η συζήτηση δεν ήταν ομόφωνη, νομίζω όμω ότι θα πρέπει να δούμε ότι τα θέματα ασφάλεια είναι θέματα κρατικά, είναι θέματα των κρατών μελών. Η πλήρη, το να πληρούνται οι προποθέσει δεν έχει να κάνει με του τους επιβάτε. Ένα όμω αν όμω γίνει ένα ε, ατύχημα, τότε ναι, αυτό φυσικά πλήττει άμεσα τους ε, επιβάτες. Ε, αυτά προς το παρόν από μένα. Ένα πολύ σύντομο σημείο ακόμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι επιβάτες ε, στο τέλος να έχουν ε, και ασφάλεια ε, των τιμών που πληρώνουν. Θα πρέπει από νωρί να ξέρουν ποια είναι η τελική τιμή των εισιτηρίων τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το συζητήσουμε και κυρίως να δούμε πώς κλείνουν τα εισιτήρια online. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να ρίξουμε περισσότερο φως. Ο συνάδελφος λοιπόν θα έρθει σε λίγο, οπότε θα σας αναφέρει και αυτός παραπάνω τα σχόλιά του. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μπράντμπορν, για την ευαισθησία που δείχνει. Προτείνει αυτή την γνωμοδότηση, αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, όπου υπάρχει αρκετή συνένεση, γιατί άκουσε τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών, των πολιτικών ομάδων, τόσο ώστε να λάβει υπόψη τις απόψεις τους και να απαλύνει τις διαφορές που υπήρχαν. Νομίζω λοιπόν ότι το κείμενο που προτείνει είναι, το κείμενο αφετηρίας προτείνει είναι καλό, καλή βάση. Ίσως το σημείο το οποίο δημιουργεί τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι αυτός ο ορισμός των περιφερειακών αεροδρομίων. Γιατί ο ορισμός μας, ορισμός μας είναι αρνητικός. Δεν μπόρεσαμε να βρούμε, δεν μπόρεσε ο εισηγητής να βρει έναν ορισμό θετικό. Μάλιστα, ο ορισμός των περιφερειακών αεροδρομίων είναι ακριβώς αυτά τα αεροδρόμια, αεροδρόμια που δεν είναι τα κεντρικά, τα κομβικά, που δεν είναι hubs. Ε, νομίζω που δεν είναι αρνητικός ορισμός. Όλοι μαζί θα πρέπει να βρούμε έναν ορισμό ο οποίος να είναι θετικός. Ποια είναι, όχι ποια δεν είναι. Επίσης ο εισηγητής λέει ότι ο ορισμός χρησιμοποιείται μόνο και μόνο στα πλαίσια της έκθεσης. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να διακρίνουμε και άρα να μην συμπεριλάβουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση αυτά τα αεροδρόμια τα οποία παρότι δεν βρίσκονται στην πρωτεύουσα μιας χώρας δεν έχουν προβλήματα εσόδων. Υπάρχουν πολλά αεροδρόμια που δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε περιφερειακά, γιατί περνάει τόση, τόση κίνηση από εκεί, υπάρχει τέτοια ροή, που τα έσοδά του, οι πόροι του είναι μεγάλοι. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν ορισμό πάλι που να λαμβάνει υπόψη αυτό το σημείο. Επίσης, η παράγραφος 1 είναι θετική. Ζητάει να υπάρχει αυτή η υποχρέωση παροχής υπηρεσίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτήν την παράγραφο, να μπει και να εκτιμώντας που να λέει ότι τα πραγματικά αυτά περιφερειακά ευρώμικα είναι σημαντικά για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις μορφές της. Και συχνά είναι η μόνη διασύνδεση ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, εδαφική συνέχεια όλων αυτών των περιοχών, ειδικά των νησιών και των, περι... απομακρυσμένων περιοχών που έχουν διαφορετικά προβλήματα σημαντικής φύσεως. Τώρα, στο σημείο που μιλάμε για το περιβάλλον και την καινοτομία δεν υπάρχει μια αναφορά στους τρόπους κατασκευής των μελλοντικών αεροδρομίων. Θα μπορούσαμε λοιπόν εδώ να βάλουμε μια τροπολογία για να ευαισθητοποιήσουμε τους θεσμικούς παράγοντες και να λάβουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς, εδαφικούς και γεωλογικούς παράγοντες τη στιγμή που αποφασίζουν πού θα χτίσουν τα αεροδρόμια. Επίσης, υπάρχει ένα σημείο που μοιάζει να είναι εκτός θέματος, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Γιατί αποκτά και μεγαλύτερη σημασία. Μία τροπολογία για την ποιότητα της εργασίας στα αεροδρόμια και την ποιότητα, τους, την ποιότητα της εργασίας που ζητάμε από τους παρόχους υπηρεσιών. Ε, μπορούν, υποτίθεται λέμε, να λειτουργήσουν ως ε, καταλήτες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αλλά θα πρέπει αυτές τις θέσεις εργασίας να πληρούν κάποια στάνταρτ. Επίσης, ε, στην παράγραφο 9 θα πρέπει να διαβρύνουμε αυτήν την παράγραφο και να μιλήσουμε για την σύνδεση αεροδρομίων και σιδηροδρόμων Ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε το δυναμικό αυτών των αεροδρομίων όλη η εμπειρία που έχουν οι, οι συνάδελφοι από τις πτήσεις ε, σε περιφερειακά αεροδρόμια μπορεί να είναι υποφελής ούτω ώστε να βελτιώσουμε την εκθεσή μας και να αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία. Πιστεύω ότι όλοι μας στα αεροδρόμια αυτά βλέπουμε ποια είναι τα όρια τους. Παραδείγματο χάρη, ε, όσοι έχουν ε, προβλήματα κινητικά και γενικά κάποιες αναπηρίες. Ε, θα πρέπει να πούμε, ε, να αναφέρουμε τέτοιου τύπου συγκεκριμένα σχόλια. Αυτά πρώτα και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Από τους πράσινους. Ευχαριστώ. Καταρχά ευχαριστώ τον συνάδελφο Bradburn για την ε, πολύ καλή συζήτηση που κάναμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία που είχαμε. Κάποια σημεία Βεβαίω θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Βεβαίως ε, δεν νομίζω ότι θα λάβουν ε, μεγάλη πλειοψηφία, παρόλο που είναι σημαντικά. Ένα το είπε ήδη ο συνάδελφος, το θέμα της διαφάνειας. Ήδη μιλούμε για τα ε, περιφερειακά αεροδρόμια για τα οποία έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα με κρυμμένες επιδοτήσεις όπου μιλούμε πάντα για το ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείες κυρίως από την Ιρλανδία για τα αεροδρόμια τους απαιτούν να, τους, ε, να υπάρξουν επιδοτήσεις. Ε, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένας τρόπος που τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Οπότε εδώ χρειάζεται σημαντική αύξηση της ε, διαφάνειας γιατί από αυτό εξαρτώνται πολλά. Γιατί αυτή η συγκέντρωση στους, ε, στις εταιρείε χαμηλού κόστους για κάποια αεροδρόμια δημιουργεί ε, κάποιες ε, θέσεις εργασίας ή κάποιες δομές εργασίας οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Δεύτερο σημείο. Ο ορισμός. Τι είναι τελικά ένα περιφερειακό αεροδρόμιο. Έχουμε διάφορες, ε, έτσι, διάφορες περιπτώσεις. Τα αεροδρόμια ας πούμε, που έχουν μεγάλη α, κίνηση, εποχιακή κίνηση, α, ε, αεροδρόμια που βρίσκονται σε ε, προορισμούς διακοπών. Α, αυτά νομίζω ότι ναι, δεν θα πρέπει να είναι τα περιφερειακά αεροδρόμια που στα ορίζουμε, τα οποία βρίσκονται σε μεγάλες πρωτεύουσες χωρών. Εδώ θα χρειαστεί συντονισμός και θα χρειαστεί και συνεργασία με, άλλες, με, άλλα μέσα ε, μεταφοράς. Να υπάρξει δηλαδή η διασύνδεση των διαφόρων ε, τρόπων μεταφοράς. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πιο σοβαρά υπόψη στην έκθεση. Επίσης, κάτι άλλο που θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό είναι ε, να υπάρξει έτσι μία άποψη για την διασυνοριακή συνεργασία. Ε, υπάρχουν ε, πολλά αεροδρόμια που βρίσκονται σε σύνορα κοντά, αλλά η σύνδεση με το επόμενο γειτονικό κράτος ας πούμε ε, δεν υπάρχει. Ε, Αυστρία, Σλοβακία, Γαλλία, Ισπανία, ε, όλα αυτά τα προβλήματα προκύπτουν σε τέτοιες οριακές, συνοριακές μάλλον περιοχές. Η σύνδεση υπάρχει μέχρι ένα σημείο αλλά από εκεί και πέρα η διασυνοριακή σύνδεση λείπει. Νομίζω ότι αυτό το σημείο στην έκθεσή σας θα πρέπει να το διευρύνετε συμπεριλαμβάνοντας και αυτό. Και επίσης νομίζω ότι η προσφορά που υπάρχει και οι πληροφορίες που δίνονται για τη σύνδεση με τα περιφερειακά δίκτυα μεταφορών ή, για, ή με τα ε, δίκτυα, με, τις, με τους τρόπους μεταφοράς που μειώνουν την ε, μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ε, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Επίσης, η τουριστική περίοδος που είναι ιδιαίτερως επιβαρυντική και ειδικά σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις των αποσκευών. Αυτό είναι ένα θέμα ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών που είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η συγκέντρωση τουρισμών είναι σίγουρο ότι είναι δύσκολο να αποφευθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αφού δεν υπάρχουν τσέχικα ή σλοβάκικα, πρέπει να χρησιμοποιήσω τις άλλες γλώσσες. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά άλλες γλώσσες δεν ξέρω. Αυτή είναι μια σημαντική έκθεση. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια πτώση των αεροπορικών μεταφορών. Σε όλη την Ευρώπη σχεδόν. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που εντοπίζω. Δεν υπάρχει συντονισμός με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με την Κίνα, Φερρυπή σε ό,τι αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις. Αυτοί δίνουν τεράστιες επιδοτήσεις. Ε, δεν ξέρω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Το θέμα δεν αφορά μόνο τα περιφερειακά αεροδρόμια, αφορά όλα τα αεροδρόμια. Επίσης, οι συνθήκες εργασίας. Ειδικά στα περιφερειακά αεροδρόμια, είναι από το κακό στο χειρότερο. Πάντα υπάρχουν προβλήματα, γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι μάλλον κακές. Το επόμενο πρόβλημα υπάρχει στον ορισμό των περιφερειακών αεροδρομίων. Δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος δυνατός ορισμός. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Επίσης για την συνδεσιμότητα. είναι περιφερειακό πρόβλημα. Το ανέφερε και ο κύριος Σουτζίας. Επίσης είναι σημαντικό να αυξήσουμε την ασφάλεια. Δεν πιστεύω όμως ότι η ασφάλεια του αεροδρομίου θα πρέπει να πληρώνεται από τις, τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Δεν το κάνουμε στις άλλες μεταφορές αυτό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις αεροπορικές μεταφορές ε, ισότιμα. Θα πρέπει να υπάρχει ομοφο... Ε, διαφάνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε κύριε Κόλτσεκ, ε, έχουμε μικρή αίθουσα, γι' αυτό δεν έχουμε πλήρη διερμηνία. Αλλά δεν είναι σωστό η Επιτροπή Μεταφορά να έχει πάντα τις μικρότερες αίθουσες συνεδριάσεων. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Τελειώσαμε τους κοιόδης. Οι υπόλοιποι θέλω ε, να μιλήσουν για δύο λεπτά. Ο κύριος Κούν πρώτος παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονικό όριο. Ευχαριστώ τον κύριο Bradburn που ανέβαλε το θέμα αυτό, την έκθεση αυτή τη ίδια πρωτοβουλία για τα περιφερειακά αεροδρόμια, γιατί όντω τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη των φτωχών σε υποδομέ περιφερειών. Οι ιδιοκτήτε αυτών των αυτών των ιδιοκτητών είναι οι πόλεις, είναι οι περιφέρειες και θα πρέπει να διατηρήσουν την, τις, τις υποδομές έτσι όπως είναι οι υποδομές αντίστοιχα στις, στα μεγάλα αεροδρόμια. Δεν μπορούν να κάνουν ε, μειώσεις, οπότε πρέπει να δούμε τι συμβαίνει για, τις, για τα μεγάλα αεροδρόμια και επίσης πρέπει να δούμε όντως τον ορισμό των ε, μεγάλων, ε, των ε, περιφερειακών συγγνώμη, αεροδρομίων. Γιατί αυτό είναι θέμα ύπαρξης για τις περιφέρειες αυτές. Θέλουν να υπάρχουν μεγάλη, μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία που έχουν charter πτήσεις για να έχουν τουριστική ροή. Και αυτό θα είναι δυνατό μόνο και αν μπορέσουμε να, πληρω... να συμπεριλάβουμε σε όλο αυτό και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε βεβαίω πρέπει να καταβάλουν και τα απαραίτητα τέλη Κάτι που πολλέ φορέ δεν συμβαίνει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με τα περιφερειακά αεροδρόμια. Εμεί είμαστε Επιτροπή Μεταφορών αλλά και υπεύθυνοι για τον τουρισμό και για την οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα των περιφερειακών αεροδρομίων πρέπει να το δούμε και να βρούμε τελικά ε, πρακτικέ λύσει. Η κυρία Φώστερ, δύο λεπτά. Yeah, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω την έκθεση Bradburn. Είναι επίκαιρη στιγμή να θέσουμε αυτά τα θέματα ξανά. Είναι πολύ σημαντικό στο γενικό πλαίσιο να... Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει πίεση για τα κεντρικά κομβικά αεροδρόμια ε, και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία των περιφερειακών αεροδρομίων. Άκουσα πολλά σχόλια για τον ορισμό. Προσπαθεί να απλουστεύσει. Ούτω ή άλλω ένα διεθνή ορισμό ε, δεν υπάρχει και προσπαθεί ο κ. Μπράντμπορν να δώσει ένα απλό ορισμό. Συμφωνώ με αυτό το θέμα της μίας, της μίας Υπάρχουν αεροδρόμια που έχουν κρατήσει αυτόν τον κανόνα. Ε, μετά τις ε, τρομοκρατικές απόπειρες. Όλοι σχεδόν είχαν δεχτεί αυτόν τον κανόνα. Ε, αυτό δεν είναι θέμα αεροπορικής εταιρείας. Αν, σας παρακαλώ μην μιλάτε, ότι πρέπει να υπάρχει μία αποσκευή στο αεροπλάνο, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά άλλο θέμα είναι ε, αυτό της μίας αποσκευής στο αεροδρόμιο. Για το, τη χρέωση των, στην πιστοτική κάρτα. Μερικές ε, χρεώσεις είναι ληστρικές. Το θέμα της διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω πάντως ότι η έκθεση Bradburn είναι σφαιρική, είναι πλήρης, έχει καλύψει τα πάντα και είναι καλή χρονική στιγμή για να θέσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ο, ο κύριος Σασόλη έχει φτάσει και του δίνω το λόγο. Δύο λεφτά όμω, κύριε Σασόλη, έτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Σιγητά, κύριε Bradburn. Αλλά συχνά η κοινοβουλευτική μας οργάνωση είναι αναποτελεσματική και δεν μας επιτρέπει να φτάσουμε στην ώρα μας. Συμφωνώ, ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα πιο σαφή ορισμό των περιφερειακών αεροδρομίων, ούτω ώστε να μην υπάρχουν αμφισημίες. Φερρυπίν στην Ιταλία. Θα ήταν να, αστείο, γελίο να θεωρήσουμε τη Μαλπένσα, το αεροδρόμιο του Μιλάνου, να θεωρήσουμε ότι είναι περιφερειακό. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε περιφερειακό κάθε αεροδρόμιο που δεν είναι hub. Που δεν είναι κομβικό, δηλαδή κεντρικό. Για τις κρατικές ε, ενισχύσεις. Συχνά η χρηματοδότηση σε αυτά τα αεροδρόμια είναι σημαντικά για την ανάπτυξη αυτού του αεροδρομίου και την ανάπτυξη της περιφέρειας που βρίσκονται. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να ανταποκρίνονται ε, αυτές οι ενισχύσεις στους κανόνες, Τα μην υπάρχουν καταχρήσεις. Υπάρχουν προσανατολισμοί ήδη από την Κομισιόν. Και παρόλα αυτά όμως συχνά αγνοούνται. Θα πρέπει οι δημόσιες αυτές ε, ενισχύσεις να μην γίνουν μια μορφή εκβιασμού στα χέρια των ε, αεροπορικών εταιριών. και να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα λεφτά, ας πούμε, απέναντι στους α, ε, δημόσιους φορείς για να πούνε θα πάμε στην τάδε περιοχή και όχι στη δίνα περιοχή. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ξανά τους κανόνες για την, ε, μία αποσκευ... την ενιαία αποσκευή και τους κανόνες για τη χειραποσκευή. Θα πρέπει να είναι ισορροπημένοι αυτοί οι κανόνες. Και δεν θα πρέπει να δημιουργούν πρόβλημα στις ε, λιανικές πωλήσει που είναι σημαντική πηγή εσόδων για τα αεροδρόμια. Επίσης, Νομίζω ότι αν υπάρχει ε, συντονισμός για τις χρονοθυρίδες μπορούμε να αυξήσουμε την ε, αποτελεσματικότητα των αεροδρομίων. Επίσης, το βασικό ενός τέτοιου αεροδρομίου είναι ότι εξυπηρετεί μία περιφέρεια. Όταν ε, συχνά σήμερα δεν υπάρχει σωστό δίκτυο μεταφορών. Επίσης, οι περισσότερες πτήσεις, τελευταία παρατήρηση, από και προς τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι από εταιρείε low cost. Ε, και επίσης έχουμε την αρχική τιμή ας πούμε, του εισιτηρίου και μετά προσθέτουμε υπερβολικά πολλές χρεώσεις έξτρα. Επίσης, πολλές υπερχρεώσεις στις επιστοτικές κάρτες. Θα, πρέπει να θεωρηθούν αυτά α, παράνομες χρεώσεις και θα πρέπει να υπάρξει κοινοτική νομοθεσία. Ας πούμε, η Ryanair ε, βάζει 2 ευρώ επιπλέον ε, για θέματα που θα πρέπει να πληρώσει η ίδια. Σε κάθε εισιτήριο ισχύει αυτό. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή δουλειά του. Και sulla... Ο Φιντάντσα. Επίσης, για τον ορισμό συμφωνώ με τον κύριο Ουτζίας και τον κύριο Σασόλη για, τις, ε, για τα περιφερειακά, τα μη hub δηλαδή, έχουμε μια μεγάλη ποικιλία αεροδρομίων. Θα πρέπει μέσω τροπολογιών που θα υποβάλουμε τις επόμενες μέρες να βρούμε έναν καταλληλότερο ορισμό για να λάβει υπόψη αυτή την πλειάδα των non-hub αεροδρομίων. Επίσης, θα πρέπει να δούμε... Θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια που είναι πολύ σημαντικά για την πολιτική την εδαφική αλλά και την πολιτική, την τουριστική της Ευρώπης. Ε, επομένως, η έμφαση που θα δώσουμε ε, σε αυτό το θέμα έχει πολλές επιπτώσεις. Κυρία Λίχτεμπέργκερ, ε, αναφερθήκατε στη Βόρεια Ιταλία. Τη γνωρίζω αρκετά καλά αυτήν την περιοχή. Εμείς έχουμε έναν φοβερό πολλαπλασιασμό αεροδρομίων εκεί. Συχνά δεν μπορούν να επιβιώσουν. παρά μόνο χάρη στις δημόσιες επιδοτήσεις από τους δημόσιους φορείς κτλ. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίκτυο μικρών αναδρομίων να, να το εξορθολογήσουμε. Και κάθε ένα από αυτά θα πρέπει, ας πούμε, αν θέλετε, να έχει το δικό του ρόλο και τη δική του αποστολή. Και κάποια να τα κλείσουμε ενδεχομένω όταν δεν καταφέρουν να επιβιώσουν στην αγορά. Ειδικά σε... σήμερα, όταν ε, ζούμε αυτή την κρίση και όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ε, πολλά δημόσια κονδύλια και οι τοπικές αρχέ δεν έχουν πολλά κονδύλια, θα πρέπει να δούμε αυτή την ιστορία. Επίσης, συμφωνώ με όλα όσα άκουσα. Πριν από λίγες μέρες διάβασα ότι ο Επίτροπος Κάλλας ε, απαντώντας ε, σε μία ερώτηση για τις υπερχρεώσεις ε, στις πιστοτικές κάρτες που επιβάλλουν κάποιες εταιρείες, είπε ότι θέλει η Κομισιόν να παρέμβει για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο της υπερχρέωσης. Θέλουμε και εμείς να πιέσουμε την Κομισιόν, ούτω ώστε αυτό το πρόβλημα να επιληθεί πάρα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκράμερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Τα περισσότερα ε, περιφερειακά αεροδρόμια βεβαίως ε, έχουν να κάνουν με το πρεστής κυρίω της ε, περιοχής. ξέρουμε ότι δεν, οι αεροπορικές εταιρείε δεν ε, επιβάλλουν νέα νέες τιμές για την ε, κυροζήνη. Ε, ξέρουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν στην Γερμανία δύο ε, πόλεις που είναι 30 χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη. Έχουν και δύο αεροδρόμιο, δεν έχουν εθνικό συντονισμό, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό συντονισμό, υπάρχει μόνο το, το σύνορο μεταξύ των κρατηδίων. Και τα δύο αυτά αεροδρόμια δεν συνδέονται. Ε, και επιδοτούνται ε, ξεχωριστά και τα δύο. Ζητούν συνέχεια ε, χιλιάδες εισιτήρια και τελικά αγοράζονται τα ελάχιστα από όλα αυτά. Το θέμα λοιπόν είναι απλώς το πρεστή της περιφέρειας. Τα, τα περιφερειακά αεροδρόμια ούτως ή άλλως δεν έχουν άμεσες πτήσεις. Πρέπει κανείς να περάσει από αυτά για να α, πάει στον τελικό του προορισμό. Σήμερα μόλις 10 α, σιδηροδρομικές γραμμές υπάρχουν, 10 ε, τρένα πηγαίνουν στο αεροδρόμιο στο Βραδεμβούργο, ενώ παλιά ήταν 100. Προφανώς οι ε, αεροπορικές εταιρείε έχουν ε, κλέψει την παράσταση σε αυτό, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Πρέπει λοιπόν τα πράγματα να αλλάξουν. Αλλιώς τα πράγματα είναι άχρηστα στην, ας πούμε, στην πολιτική για τους σιδηροδρόμους στην Γερμανία τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσει. Οι ε, αριθμοί των επιβατών μειώθηκαν κατά 20%. Η περιφερειακή ε, ε, μετακίνηση λοιπόν αυξήθηκε κατά 50%. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Γιατί αλλιώ 90% των περιφερειακών αεροδρομίων θα πτωχεύσουν. Η Κομισιόν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι είστε πιεσμένοι από χρόνο. Θα είμαι λοιπόν λακωνικός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί την έκθεση Bradburn δίνει τροφή για σκέψη και συμβάλλει σημαντικά σε αυτή τη συζήτηση. Θα την εξετάσουμε δελεχώς τι επόμενες εβδομάδες. Και συμφωνούμε με το μου ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια θα διαδραματίσουν σωτικό ρόλο στην εδαφική ε, συνοχή και στην καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των περιφερειών και θα αποσυμφορήσουν τα πολύ ε, γεμάτα κομβικά αεροδρόμια. Τώρα, τα περιφερειακά αεροδρόμια δεν έχουν κομβική λειτουργία. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να περιληφθούν σε ένα περιεκτικό δίκτυο γιατί εξυπηρετούν κυρίως ε, περιφερειακές ανάγκες. Ε, βέβαια, θα συνδέονται με τα κομβικά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, περιλαμβάνονται στο βασικό δίκτυο. Γιατί είναι αυτή η προσέγγιση μας, γιατί πιστεύουμε ότι και οι σιδηροδρομικές ε, διασυνδέσεις ε, είναι αποτελεσματικές όταν υπάρχει μια ελάχιστη συγκέντρωση σε συγκεκριμένο δρομολόγιο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Βέβαια, γι' αυτό έχουμε και τόσο ακριβέ υπερταχίες που ουσιαστικά αντικαθιστούν τις αεροπορικές μεταφορές σε πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό ε, ορίσαμε ένα ελάχιστο κατόφλι για τα κεντρικά, τα κομβικά αεροδρόμια. Τώρα για το θέμα της ε, διατροπικότητας. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μας και ήδη εκπονούμε έναν οδικό χάρτη προκειμένου να υποβάλουμε και μια οδηγία για την ε, ενιαία έκδοση εισιτηρίων ε, που βρίσκεται στην καρδιά της πρότασής μας για την πολυτροπικότητα και την, το ενιαίο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Επίσης, ε, έχουμε και μια ειδική ομάδα εργασία ε, που εξετάζει τη συμβολή της διατροπικότητα ε, για την αποσυμφόρηση, την καλύτερη προσπελασιμότητα και τα υπερβολικά επίπεδα προσαρμογής. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των τιμών, που επισημάνθηκε από πολλούς ομιλητές, είναι σημαντικό το θέμα της διαφάνειας, γιατί κάποιες low cost κυρίως αεροπορικές έχουν την τάση να επιβάλλουν σχεδόν αναπόφευκτα επιπλέον χρεώσεις ε, επί της βασικής τιμής δηλαδή. Αναφέρθηκε ε, το θέμα το, της χρήσης πιστοτικών και χρεωστικών καρτών, ειδικών. Ε, είναι, αρχίζει και αποκτά διαστάσεις. Ήδη θα αναθέσαμε μια εξωτερική μελέτη για τέτοια θέματα με βάση τον κανονισμό ε, 1008 και 2008 και υπάρχουν διαφορές στον τρόπο πληρωμής αλλά ε, θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να ε, υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης επιλογής πληρωμής, κάτι που δεν ισχύει πάντα. Θα το αντιμετωπίσουμε φέτος ε, με τις ρυθμιστικές αρχές στα κράτη-μέλη για να δούμε τι θα επιτρέπεται και τι όχι δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας και τι συμπεράσματα θα αντιλήσουμε από την κατάσταση αυτή. Και τέλος, για, για τον περίφημο κανόνα της μίας και μόνη αποσκευής. Θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των συμφερόντων των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων και των συμφερόντων των επιβατών. Αν δούμε τις συνέπειες αυτών των πολιτικών στις πωλήσει ελληνικού εμπορίου στα ε, αεροδρόμια, βλέπουμε ότι είναι θέμα ε, business to business μεταξύ των αερολιμένων, των αεροπορικών εταιριών, δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων. Οπότε, μια και πρόκειται για θέματα ανταγωνιστικότητας, εμπίπτει σε θέματα ε, νομοθετικών διατάξεων περί ανταγωνιστικότητα. Δεν χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία. Γιατί το νομοθέτημα αυτό στόχο έχει την προστασία των, των καταναλωτών, την προστασία των επιβατών. Σε ό,τι αφορά τώρα του επιβάτε. Όντω, κάποιοι επιβάτες ε, μπερδεύτηκαν από τους πολυάριθμους περιορισμούς που ισχύουν για την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών από προσωπικό εδάφους στους αερολιμένες. Βέβαια, εξετάζουμε αυτό το θέμα των αποσκευών και χειραποσκευών για να δούμε τι θα γίνει με τον κανονισμό 261 ε, που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Και μάλιστα πρόσφατα ξεκινήσαμε δημόσιες διαβουλεύσεις προκειμένου να καλέσουμε τους ενδιαφερόμενους να συμβάλλουν με προτάσεις ε, και πιθανές λύσεις για τα θέματα αυτά των αποσκευών και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι πρακτικές ε, των ε, αγορών σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, εισφορές, τις επιπλέον, δαπάνε δαπάνες για τις αποσκευές ή τις χρεώσεις για τις αποσκευές. Ο κύριος Μπράντμπον, ο εισηγητής μας, για να ολοκληρώσει. Θα ήθελα εν συντομία να απαντήσω σε ορισμένα σχόλια των συναδέλφων. Οι παρατηρήσεις ε, μίλησαν, ε, ε, οι παρατηρήσεις επικεντρώθηκαν σε σημαντικά θέματα. Ο κύριος με ο κύριος Ουτζίας μίλησαν για τις αποσκευές, για τα θέματα της ασφάλειας. Είναι κεντρικά ζητήματα της έκθεσης και επανερχόμαστε σε ένα ζήτημα που ήδη απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις πιο τα πιο αυστηρά μέτρα. Δεν είναι θέματα γενικής ασφάλειας, ε, γενικών διατάξεων ασφάλειας, αλλά πιο αυστηρών μέτρων. Και η έκθεση το αναφέρει. Το θέμα του ορισμού των περιφερειακών αερολιμένων. Κάποιοι συνάδελφοι <clears throat> επισήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις δικές τους πατρίδες. Βέβαια, πολλά από αυτά ε, σχετίζονται με τις ε, εθνικές πολιτικές. Ο κύριος Φιντάντσε και ο κύριος Ασόλη μίλησαν για την ε, υποβάθμιση που έκανε η τελική κυβέρνηση του αεροδρομίου του Μιλάνου, της Μαλπέσα, που το χαρακτήρισε περιφερειακό. Αυτό δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν έχουμε ένα κοινοτικό ορισμό, ε, δεν θα εμπίπτει πια αυτό το θέμα ο χαρακτηρισμός σε εθνική πολιτική. Το ζήτημα της διαφάνειας επίσης ε, αναφέρθηκε από πολλούς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για εμπορικές ε, δραστηριότητες και ισχύει και ο ανταγωνισμό. Σωστό αυτό. Αλλά τι γίνεται με τον καταναλωτή, γιατί ο επιβάτης, ο καταναλωτή στερείται πληροφοριών ε, πριν φτάσει στο αεροδρόμιο εξαιτία ε, της πληθώρας των αερογραμμών, των αεροπορικών εταιριών. Και όταν κανείς κάνει κράτηση του εισιτηρίου δεν ξέρει πόσο ουσιαστικά θα πληρώσει, πόσο θα χρεωθεί η αποσκευή του και ενώ υπολογίζει σε μια βασική τιμή βλέπει ότι πληρώνει 30-40 ευρώ επιπλέον για τις αποσκευές. Σίγουρα στηρίζουμε την εμπορική δραστηριότητα, αλλά χρειαζόμαστε και διαφάνεια για τους επιβάτες. Το ίδιο ισχύει και για τις χρεώσεις των πιστοτικών καρτών. Κύριε Χίγκης, με κάθε σεβασμό δεν νομίζω ότι κανένας είπε ότι, δεν, ότι απαγορεύεται η χρέωση για τη χρήση πιστοτικών καρτών, αλλά θα πρέπει να είναι λογική αυτή η, η χρέωση και όχι υπερβολική και καταχρηστική εκ μέρους των αεροπορικών εταιριών. Γιατί μερικές φορές είναι υπερβολικέ οι χρεώσει εκ μέρους των αεροπορικών εταιριών. Ξεπερνούν κατά πολύ το κόστος ή τι δαπάνε του ντοσιέ. Θέλουμε λοιπόν μία λογική χρέωση με βάση το κόστος ε, που καταβάλει ο αερομεταφορέας. Ένα άλλο σχόλιο κύριε Πρόεδρε αφορά το ζήτημα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και του βασικού δικτύου Core Network. Αυτό που λέμε στην έκθεση δεν είναι ότι κάθε αεροδρομιάκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περιληφθεί στο, στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αλλά εφόσον εξυπηρετεί ένα αεροδρόμιο σημαντικές και μεγάλες περιφέρειες και μπορεί να συμβάλλει ε, στην βελτίωση των αεροπορικών μεταφορών και να τις ενισχύσει, τότε μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο δεν ε, θα πρέπει μόνο τα κομβικά αεροδρόμια να περιλαμβάνονται σε διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, γιατί και περιφερειακά αεροδρόμια έχουν τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό και θα πρέπει να τα εξετάσουμε περιπτωσιολογικά το κατά πόσο θα συμπεριληφθούν ή όχι στα TEN, στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτά, Πρόεδρε, και προσβλέπω στη συνέχεια τη συζήτηση ε, με την πορεία ε, τη έκθεση μου. Ευχαριστώ, κύριε Μπράτμορ. Να σα υπενθυμίσω ότι η διορία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση Μπράντμπορν ε, είναι η 3η Φεβρουαρίου. Θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο στην Επιτροπή Μεταφορών και έχει προβλεφθεί η έκθεση για την δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Λοιπόν, η διορία για τις τροπολογίες η 3η Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν και περιμένουμε και κλείνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Κάλλας. Αρχικά προβλεπόταν ανταλλαγή απόψεων για το πακέτο για τους αερολιμένες, αλλά μετά το τραγικό ναυάγιο στις ακτές Ιταλίας με το κρουαζιερόπλιο Κονκόρντια ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από τον κύριο Κάλλας να μας κάνει μια δήλωση και μια ενημέρωση για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ως εκ τούτου το πρώτο ημίωρο της συζήτησης ε, με τον Επίτροπο θα αφιερωθεί στο ναυάγιο του κουραζιερόπλου Κονκόρδια. Παρακαλώ λοιπόν κύριε Επιτροπέ, έχετε την καλοσύνη να μας ενημερώσετε για τις τελευταίες εξελίξεις ως προς το Κονκόρδια. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε για ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μετά το ναυάγιο του Κώστα Κονκόρδια. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα θύματα. Έστειλα επιστολή στον Ιταλό Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κόνραντο Πανσέρα, για να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για το τραγικό αυτό ναυάγιο και τα θύματα. Και φυσικά παρισχά την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλισης για να συμμετέχουμε σε, σε σωστικές επιχειρήσεις οι σωστικές αυτές επιχειρήσεις ε, συνεχίζονται και γίνονται προσπάθειες για να αφαιρεθούν ε, πάνω από 2.300 τόνοι πετρελαίου που βρίσκονται στο πλοίο για να αποφευθεί ε, ο κίνδυνος πετρελοκυλίδας. Επίσης, έχει δοθεί από τον ΟΗΕ ένα ειδικό σκάφος που βρίσκεται σε επιφυλακή υπό την αιγίδα μιας ειδικής επιχειρήσεις διάσωσης. Και περιμένουμε εξελίξεις γιατί όλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα ε, προκειμένου να ξεκινήσει η άντληση του πετρελαίου από το Κροσγερόπουλιο, που αναμένεται να ξεκινήσει ανα πάσα στιγμή. Τώρα, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς εμπλέκονται όλοι αυτοί και πώς παρακολουθούν την υπόθεση. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση, εξετάζουμε την νομοθεσία μας, προσπαθούμε να βρούμε κάποιες αδυναμίες αν υπάρχουν, αλλά πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι και λογικοί. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι το υπαριθμό ένα ζητούμενο. Και έχουμε ταυτόχρονα δύο παράλληλες διαδικασίες. Η μία αφορά τις έρευνες για το ναυάγιο και το δυστύχημα του Κώστα Κονκόρδια και έχουμε τακτικές και συνεχείς επαφές με τις Ιταλικές αρχές, τις οποίες ήθελα να ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία που μας παρήχαν. Και όταν ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή για το δυστύχημα του Κώστα Κονκόρδια, θα κάνουμε μια αξιολόγηση των συμπερασμάτων και θα αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση του Κουρασγερόπουλου Κώστα Κονκόρδια. Η δεύτερη παράλληλη διαδικασία είναι το τακτικό μας έργο της ενημέρωσης επικαιροποίηση των προδιαγραφών ασφάλειας στην αυσιπλοεία και για ασφάλειας και των επιβατών και των πλοίων. Ασφάλεια επιβατών, ασφάλεια πλοίων και αποφυγή της ρήπανσης. Έχουμε και ευρωπαϊκά και διεθνή αρμόδια όργανα. Η ναυσιπλοεία είναι μια παγκόσμια οργάνωση, γι' αυτό και έχουμε και τη Διεθνή Οργάνωση για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς συμβάλλει στην νομοθετική διαδικασία προκειμένου να εφαρμόσει και να αναβαθμίσει τους κανόνες ασφάλειας στο μέτρο του δυνατού. Είμαστε πολύ δραστηροί, ε, θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές για την ασφάλεια. Οπότε δεν μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Δεν περιμένουμε να γίνει δυστύχημα για να αναλάβουμε δράση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις και αναθεωρήσεις πολιτικών και της σχετικής νομοθεσίας ε, για την ασφάλεια καθώς και τα προληπτικά μέτρα. Δηλαδή επιτελούμε το έργο μας. Στόχο μας είναι να ε, ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των διατάξεων ασφάλειας και για τους επιβάτες και για τα πλοία και να εφαρμόσουμε παρόμοιες προδιαγραφές για όλα τα επιβατικά πλοία που ελιμενίζονται ή αποχωρούν από κοινοτικά λιμάνια. Επίση, θέλουμε να βελτιώσουμε τη σταθερότητα των ε, επιβατικών πλοίων μετά από βλάβη του ή από σύγκρουση. Επίσης το θέμα της καταχώρηση ε, των επιβατών και ε, διαδικασία εκένωση του πλοίου είναι πολύ σημαντικά θέματα. Θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσει για να βελτιώσουμε τι προδιαγραφέ ασφάλεια των επιβατικών πλοίων. ε, τα πλοία αναπτύσσονται, η τεχνολογία εξελίσσεται, οι επιβάτες ταξιδεύουν όλο και περισσότερο, γι' αυτό θα πρέπει ε, να επικαιροποιήσουμε αντιστοίχως και τις ασφάλ... τους κανόνες ασφάλειας για τα επιβατικά πλοία. Ξεκινήσαμε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους ε, για να εξετάσουμε κάποιες λύσεις. Τα νομοθετικά μέτρα και τα συνοδευτικά μέτρα έχουν προγραμματιστεί ήδη από το καλοκαίρι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τραγικό δυστύχισμα του Κώστα Κονκόρντια, αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώ έδειξε ότι η ασφάλεια είναι το υπαριθμό ένα ζητούμενο στι μεταφορέ. Γιατί η ναυσιπλοεία έχει εντυπωσιακέ επιδόσει ασφάλεια τα τελευταία χρόνια, παρά τη τις ε, ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την ε, αύξηση των ε, πλωτών μεταφορών και των θαλάσσιων μεταφορών. Βέβαια, θα πρέπει και οι νομοθέτε να βρίσκονται σε εγρήγορση και επιφυλακή. Προσβλέπω στην υποστήριξη και του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών ε, ε, όταν θα καταθέσουμε τις μελλοντικέ μας πρωτοβουλίες προκειμένου να γίνει ακόμη πιο ασφαλή η ναυσιπλοεία. Και μάλιστα την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου, είχαμε μία συνάντηση εργασίας με θέμα τις προτάσεις ε, για την ασφάλεια των επιβατικών πλοίων. Και ο επικεφαλής εμπειρογνώμονας που είναι παρόν και σήμερα είπε ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε πριν ε, γίνει το δυστύχισμα. Πριν γίνει, να μην περιμένουμε κανένα δυστύχημα. Και αυτό ήταν στις 13 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω. Πριν το ατύχημα δηλαδή. Κύριε Επίτροπε, έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο μιλητών και πολύ περιορισμένο χρόνο. Ε, μετράω εδώ 12 ομιλητέ. Θα είμαι αυστηρό στην τήρηση του χρόνου, δύο λεπτά ο καθένα, ώστε να απαντήσει ο Επίτροπο και να επανέλθουμε στι τακτικέ μα εργασίε και στο αρχικά προβλεπόμενο θέμα τη ανταλλαγή απόψεων. Αναγνωρίζω τη σημασία του θέματο, αλλά παρακαλώ χρόνου φίδου. Ξεκινούμε με τον κύριο Φιντάντσα από το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για αυτή την ισορροπημένη και ορθολογική του προσέγγιση. Ε, στη στιγμή αυτή ε, έχουμε θέσει κάποιες προτεραιότητες. Ε, φυσικά να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες άντλησης ε, από το κουρασγερόπλιο, να ασφαλιστεί το πλοίο, να συνεχίσουμε τις σωστικές ενέργειες μήπως βρούμε πτώματα και να, και να αποφύγουμε την περιβαλλοντική καταστροφή. Αυτό είναι πιθανό γιατί από ό,τι προβλέπετε θα επιδεινωθεί ε, ο καιρός στη θάλασσα τις επόμενες μέρες και αυτό μπορεί να δυσκολέψει την ε, επιχείρηση ε, εκαθάρισης πτωμάτων κτλ. Πριν πάρουμε όμως νομοθετικές πρωτοβουλίες, θα πρέπει να περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που θα διεξαχθεί. Δεν είναι σίγουρο ότι από την έρευνα έρευνα θα, θα προκύψουν ε, προβλήματα νομοθετικών ελλείψεων κτλ. Σίγουρα θα προκύψουν ε, προβλήματα ανθρώπινου λάθους, ε, έλλειψη σωστών χειρισμών κτλ. και μη σεβασμού των κανόνων. Έχουμε ένα σύστημα κανόνων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις ε, περισσότερο, ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τις αποζημιώσεις. Ό,τι και λένε οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες, για τις ε, συνομιλίες μεταξύ καπετάνιου και λιμενικών, Υπήρχε σίγουρα ε, πρόβλημα σε ό,τι αφορά την μη τήρηση των κανόνων. Θα πρέπει να περιμένουμε ε, τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε καθήκον ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών να υποστηρίξουμε ε, με στένος ένα τομέα τουριστικό που έχει δώσει καλά αποτελέσματα και που έχει αυξηθεί και αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει και να τηρήσουμε τα, τους κανόνες ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή την εκστρατεία ε, δαιμονοποίησης, αν θέλετε, και στυλίτευσης αυτού του τομέα, ο οποίος έχει συνεισφέρει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη. Κυρία Τσερκιάνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ σήμερα. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που είπατε εσείς και σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Φιντάντζα. Θα υπάρξει μία έρευνα. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Αλλά κάτι που φαίνεται σίγουρο είναι ότι το πλοίο αυτό Κώστα Κροτσέρα έπλε πολύ κοντά στην ακτή. Μάλλον δεν είχε ακολουθήσει, μάλλον ε, αγνόησε τους κανόνες ταυσιπλοείας. Και μάλιστα αυτή ήταν μία από τις... Ε, είναι ένας βασικός κανόνας για τα κρουαζιερόπλια. Εγώ εκπροσωπώ αυτούς τους, ε, εκπροσωπώ την ομάδα των σοσιαλιστών. Και θα ήθελα να σας πω ε, για αυτό το θέμα της απόστασης από τις ακτές και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να εξασφαλίσει κάποια ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας για την ναυσιπλοεία και πρέπει να τηρούνται. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να παρέμβουμε πάρα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχουν κανόνες, ότι Και δεν πρέπει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε τους ελάχιστους κανόνες ε, ασφάλειας ε, και τους ελάχιστους κανόνες για την κατάρτιση του πληρώματος. Ε, επίσης, πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποιος θα πληρώσει τι και πόσο. Η κυρία Μάισνερ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είσαστε εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό σήμερα πρέπει, όταν προκύπτουν τέτοια θέματα, πάντα σκεφτόμαστε, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τα αποφύγουμε. Όλοι είχαμε πει ότι το Τιτανικό ήταν ένα πλοίο που δεν μπορούσε να βυθιστεί και τελικά βυθίστηκε. Θα μπορέσουμε λοιπόν ποτέ να αποφύγουμε τέτοια δυστυχήματα. Ως ε, ε, προδιαγραφές ασφάλειας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να έχουμε το μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Ε, νομίζω ότι έχουμε, φαίνεται ότι έχουμε πάρει κάποιο λάθος δρόμο. Ε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε με οποιοδήποτε, οποιοδήποτε ρύθμιση. Ε, γιατί το πρόβλημα υπάρχει, το δυστύχημα έγινε. Ένα ερώτημα λοιπόν έχω. Πολλοί λένε ότι ο καπετάνιος έκανε ε, το λάθος. Άκουσα και από ειδικού που λένε ότι ο ότι ο, ο καπετάνιος δεν έκανε κάποιο λάθος γιατί τελικά ε, απέφυγε το να ε, βυθιστεί τελειωτικά το πλοίο αφού ε, προσάραξε ουσιαστικά, στο, έγειρε πάνω στον βράχο. Ε, επίσης, ε, είπατε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει τις ε, διατάξεις για διαγραφές ασφαλείας. Επί ποιας βάσεως ο κύριος Φιντάντσα επίσης το είπε, θα πρέπει μάλλον να δούμε καταρχάς ποια ήταν η αιτία, αν τα σκεφτήκαμε όλα, αν υπήρχε κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί, τι θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον στις προδιαγραφές ασφαλείας. Υπάρχουν όλα αυτά και απλώς έγινε ένα λάθος τελικά. Τι συνέβη. Και επίσης, δυστυχώς ε, τραυματίστηκαν, ε, πέθαναν ε, επιβάτες. Θα πρέπει να Εξεταστεί λοιπόν αν όντω ε, υπήρξε ε, πλήρη στήριξη όλων των προδιαγραφών που ε, υπήρχε. Και επίση πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα δικαιώματα των επιβατών μετά από τέτοια δυστυχήματα. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Τώρα για το ποινικό τη υπόθεση, που είναι τα προβλήματα και ποιο έκανε το λάθο,. ε, ουσιαστικά πρέπει να δούμε ποιος είναι ο παράγοντας που τα υποκίνησε όλα αυτά από πίσω. Και νομίζω ότι κάποια ερωτήματα εκεί έχουν μείνει αναπάντητα. Πρώτον, συχνά βλέπουμε και ισχύει για τις, κυρίως για τις μεταφορές αγαθών, ότι Υπάρχουν ε, ε, εμπορεύματα συνήθως που υπάρχουν εμένα αλλά δεν δηλώνονται ή δεν ελέγχονται. Ερώτημα, σε αυτό, το, αυτό το φαινόμενο υπάρχει και στα μεγάλα κρουαζιερόπλια. Δεύτερο ερώτημα. Άκουσα κάποια στιγμή ότι τα, οι προδιαγραφές ασφάλειας για τα κήτη ήταν μόνο για 12 μέτρα. Ε, ναι, αλλά προφανώς αυτό ήταν μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο κροσγερόπλιο. Ισχύει αυτό και αν αυτό ισχύει νομοθετικά τι επιπτώσεις υπάρχουν. Ε, γιατί Νομίζω ότι αυτό προέκυψε από ειδικού από Γερμανία, ε, ε, Βρετανία και Ιταλία. Το πιο σημαντικό για μένα είναι το θέμα της διάσωσης, του χρόνου διάσωσης και των, και των διαθεσίμων χώρων για τη διάσωση των επιβατών, που από ό,τι φαίνεται από υπολογισμούς είχαν την ε, ε, συμπεριφορά που έπρεπε, αλλά τελικά οι πόροι που υπήρχαν δεν ε, έφτασαν για αυτούς του 4.000 ανθρώπους. Ελέγχθηκε αυτό και αν ναι, με ποιο τρόπο και από ποιον. Υπάρχουν συνέπειε κατά τον έλεγχο εφόσον προέκυψε κάτι που δεν ήταν όπως έπρεπε. Για παράδειγμα, στην, στην αεροπλοεία υπάρχουν συγκεκριμένοι χρόνοι διάσωση που πρέπει να τηρηθούν για κάποια τμήματα του αεροσκάφου, α πούμε. Κάτι τέτοιο υπάρχει Καταναλογία και στα πλοία. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Και επίσης για το πετρέλαιο αλλά και για τα υπόλοιπα χημικά στοιχεία τα οποία εκλείονται πλέον στο, στη θάλασσα. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ποιος θα πληρώσει και πώς θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Και το θέμα για την καταβολή του το κόστου. Ε, μίλησε η συνάδελφος για τον Τιτανικό. Η αποζημίωση ε, είχε υπολογιστεί τότε 100 δολάρια για κάθε νεκρό. Ε, αυτό έχει, έχει γίνει κάποιο υπολογισμό για την αποσημείωση των θυμάτων από αυτό το κροσγερόπλιο. Και ένα τελευταίο, το θέμα τη ε, εκένωση. τα σχέδια εκένωση θα ήθελα να τα ξανακοιτάξετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Okay, the list is getting longer, I'm afraid. Ο κατάλογος μακραίνει, αντί να μειώνεται. Κυρία Φώστερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν που ήρθε τόσο γρήγορα να μας μιλήσει εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Όλα αυτά που υπόθηκαν ήταν σωστά. Θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα της έρευνας του ατυχήματος. Ε, βεβαίως μπορεί να, μπορούμε να κάνουμε δίκες από τις εφημερίδες και τις, α, τις τηλεοράσεις, αλλά εμείς στην Επιτροπή Μεταφορών δεν το κάνουμε. Ό,τι και να είναι αυτό που έχει συντριβεί, που έχει πέσει κτλ, αεροπλάνο, πλοίο κτλ, περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ε, τώρα, υπήρχε το ερώτημα, πρέπει να βάλουμε περισσότερους κανόνες, δεν ξέρουμε. Ε, το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες, το θέμα είναι αν εφαρμόζονται σωστά από το πλήρωμα τη συγκεκριμένη μέρα. Δεν ξέρουμε ακόμα ε, τι προβλήματα υπήρξαν. τέθηκε το θέμα του καπετάνιου. Ε, δεν είναι μόνο ένας αξιωματικός στο πλοίο, έτσι. Ε, πολλοί έχουμε πάει από εμά σε τέτοιες ε, διακοπές σε κρουαζιερόπλοιο. Ε, φυσικά παίρνει τελική ευθύνη, ε, αλλά υπάρχουν διάφορα θέματα για τον συμπερισμό ε, των αξιωματικών. Επίσης, 4.000 ανθρώπων διασώστηκαν. Αυτό σημαίνει ότι το περισσότερο πλήρωμα έκανε θαυμάσια τη δουλειά του. Επίσης, οι Ιταλοί είναι είναι ναυτικό λαό. Ε, αυτή την τραγική στιγμή θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι οικογένειε και του αγνοούμενου. Από την δική μα πλευρά, η ΣΥΑΡ δηλαδή, περιμένουμε, περιμένουμε τι θα μας πει η Κομισιόν και όλοι οι υπόλοιποι φορείς. Νομίζω ότι στις σημερινές συνθήκες αυτό είναι το πιο σωστό να κάνουμε, να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριο Σκούν, δύο λεπτά. Από εδώ και πέρα θα είμαι αυστηρότατος. Θα τηρούμε τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Φώστερ. Όταν συμβαίνουν τέτοια δυστυχήματα, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής καταγραφή της κατάστασης. Μόνο έτσι μπορούμε ουσιαστικά να διαχειριστούμε την κατάσταση. Και αυτό είναι το πρόβλημα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Είναι το ανθρώπινο λάθος. Ε, ναι, ε, ο, ο καπετάνιος μπόρεσε να, ε, θέλησε να υποβιβάσει το γεγονός, ήταν δικό του το λάθος, ήταν καταστροφή, προσπάθησε να αποφύγει την ε, έκρηξη πανικού μέσα στο πλοίο, αλλά αν η, οι προδιαγραφές που υπήρχαν τηρήθηκαν τελικά για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. Υπάρχουν αυτά τα μεγάλα ε, κρουαζιερόπλια με τους 4 και 5.000 ανθρώπους ε, έχουν πολύ αυστηρές τέτοιες προδιαγραφές. Οι η κατάσταση αυτή λοιπόν είναι πραγματικά τραγική. Δεν υπήρχε, δεν έγινε κανένα, καμία άσκηση διάσωσης. Μήπως το, ε, το προσωπικό δεν έδωσε τις ε, εντολές για να κάνει αυτή την, αυτή την άσκηση το, το, οι επιβάτες. Δόθηκαν οι απαραίτητες εντολές. Ποια γλώσσα χρησιμοποιήθηκε. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Και τέτοια μεγάλα κρουαζιερόπλια πώς ε, να ναυπηγούνται. Και με τέτοια μεγάλα υψηλά, υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικά συστήματα και τελικά δεν υπάρχουν μέσα σε αυτό το ε, μεγάλο ε, πλοίο ούτε σωσίβια, κόβεται και το ρεύμα και ο καθένας είναι, απομένει στην τύχη του. Τι κατασκευή είναι αυτή που γίνεται σε αυτά τα τεράστια κρουαζιερόπλια. αυτά τα, αυτό το συγκεκριμένο πλοίο βρέθηκε σε μια πραγματικά τραγική κατάσταση. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, είναι σημαντικό να το δούμε. Να δούμε ποιε είναι οι προδιαγραφέ όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά και για την αφήγηση και για την κατασκευή αυτών των ε, πλοίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλιτσεκ, δύο λεπτά. Έκκληση. Δεν σας το λέω, τώρα σας κάνω απλώς έκκληση. Εντάξει, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, την επόμενη περίοδο θα εφαρμόσουμε αυτό το πακέτο για τη θάλασσα. Το έχουμε υιοθετήσει, έχουμε υιοθετήσει την οδηγία για τις α, τεχνικές έρευνες των θαλάσσιων ατυχημάτων. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εσείς, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ε, θεωρείτε ότι γίνονται σεβαστές αυτές οι οδηγίες. Είναι δυνατόν να γίνει σεβαστή αυτή η οδηγία και ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής από την, από το, τήρηση ή μη των κανόνων της οδηγίας. Δύο λεφτά. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω, κύριε Επίτροπε. Καταρχάς, για τα περιβαλλοντικά θέματα. Ορισμένα κράτη-μέλη ε, δεν θέλουν να χρησιμοποιούν αργό πετρέλαιο στα κουρασγερόπλια. Το χρησιμοποιούμε γιατί είναι πολύ φθηνό. Αλλά βλέπετε τι συμβαίνει όταν βυθίζεται το πλοίο. Υπάρχει πρόβλημα με, την, με το περιβάλλον. Δεύτερον, με τα πρότυπα ασφάλειας. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου μεγέθου πλοία που είναι ασφαλή, είναι αδύνατο να κενώσουμε ένα πλοίο με 4-5 ανθρώπου ανθρώπους πάνω. Όσο καλό και να το πλήρωμα, όσο καλή κατάρτιση και να έχει, είναι αδύνατο να κενωθεί σωστά το πλοίο. Είναι σωστό να έχουμε τόσο μεγάλα πλοία, δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο για τα κρουαζιερόπλοια. Τρίτον, δεν ήξερα ότι δεν υπάρχουν κανονισμοί γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονισμό που να λέει ότι ο καπετάνιο πρέπει να μένει πάνω στο πλοίο μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ κύριε Ουτζίας. Δύο λεπτά. Πρόεδρε. Δεν πρέπει να πούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι ιταλική. Είναι μια ευρωπαϊκή τραγωδία. Μην ξεχνάτε ότι περισσότεροι από τα θύματα δεν είναι καν Ιταλοί. Είναι Γερμανοί, είναι Γάλλοι. Ε, Θα ήθελα να εκφράσω να το πούμε αυτό. Πέρα από το ανθρώπινο λάθος, επίσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για την αξία των προσώπων. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα λάθη και ποια είναι τα όρια που έχουμε μπροστά μας. Κάτι που υπόθηκε. Υπάρχει υπερβολικός αριθμός επιβατών σε αυτά τα πλοία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Δεν μπορούμε όταν υπάρχει ε, επίγουσα ανάγκη να εκενώσουμε 4.000 άτομα σε λίγα λεφτά. Γιατί άλλο είναι τώρα να κάνουμε μια άσκηση όταν είναι το πλοίο ας πούμε ακίνητο σε οριζόντια θέση και άλλο είναι να κάνουμε άσκηση ε, που δεν είναι πια άσκηση, ε, εκένωση ουσιαστικά, όταν το πλοίο είναι σε γωνία 45 μοιρών είναι 90 μοιρών. Έπειτα, ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε συχνά ποια είναι η θέση του πλοίου, δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή τους δορυφόρους, αλλά εδώ έχει γίνει. Επίσης, πρέπει να δούμε τις πορείες των μεγάλων πλοίων μέσα από τα στοιχεία που έχουν οι λιμενικές αρχές. Δεν μπορούν οι λιμενικές ε, αρχές να προσέχουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη, ρότα του πλοίου μόνο τη στιγμή που πέφτει πάνω σε ύφαλο, ας πούμε, πάνω στις ακτές το πλοίο αυτό. Δεν γίνεται. Οι λιμενικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν αυτά τα πλοία και να εντοπίζουν νωρίς τα λάθη. Τα περισσότερα ερωτήματα ετέθησαν. Δύο σύντομα ερωτήματα θέλω να θέσω εγώ. Αναφέρατε την έμψα λίγο πριν, χωρίς να την αναφέρατε έτσι, ρητά βεβαίως υπενηχθήκατε κάτι για την ε, ΕΜΣΑ, για την ε, αλλαγή των, και την αποφυγή αυτών των δυστυχημάτων. Η ΕΜΣΑ έχει εμπλακεί όλη αυτή τη διαδικασία και αν ναι, με ποιο τρόπο. Και δεύτερον, ε, βεβαίως πρέπει να περιμένουμε την τελική έκθεση, αλλά θα με ενδιέφερε να δούμε τι γίνεται με, τα, με, την, ε, με τη σύνθεση του πληρώματος και την εκπαίδευσή του. Γιατί ίσως εκεί να υπάρχουν ε, κάποια πράγματα τα οποία να μπορούμε στο μέλλον να τα βελτιώσουμε. Ίσως και η ΕΜΣΑ θα μπορούσε στο τομέα αυτό να παίξει έναν συντονιστικό ρόλο. Σα όλοι δύο λεφτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μιλάμε για την ασφάλεια και για τα πρότυπα ασφάλειες. Μιλάμε για τις ε, έρευνες που είναι εξελίξει. εξελίξη. Το να καταλάβουμε τι συνέβη σε αυτό το πλοίο που έφερε 4.000 επιβάτες δεν είναι εύκολο, γιατί καταρχάς έσπασε το μαύρο κουτί. Μπορεί ένα τέτοιο πλοίο να ταξιδεύει με τόσους επιβάτες και μόνο με ένα ε, μαύρο κουτί. Και αν σπάσει αυτό το κουτί, αν χαλάσει δηλαδή, θα μάθουμε ποτέ τι πήγε στραβά. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι για τέτοια πλοία θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερο από ένα μαύρο κουτί. Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Δανέλης, δύο λεπτά. Νομίζω ότι πριν την ολοκλήρωση της έρευνας ε, αυτής της τραγωδίας ε, για τρία πράγματα μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Το πρώτο, ότι ενώ κανονισμοί υπάρχουν, προκύπτει το ζήτημα αν εφαρμόζονται αυτοί οι κανονισμοί και πώς ελέγχουμε την εφαρμογή των κανονισμών αυτών ώστε να προβλέψουμε παρόμοια δυστυχήματα. Το δεύτερο θέμα νομίζω ότι είναι ότι ε, είναι φανερό ότι πρέπει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των ναυτικών από την ε, απίστευτα ανάρμοστη, την απίστευτη συμπεριφορά του καπετάνιου μέχρι την επάρκεια του προσωπικού στην ε, διάσωση και τη βελτίωση των προσπαθειών αυτών. Και το τρίτο, νομίζω ότι δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε ότι τα νέα γενιά κουραζιερόπλια, με αυτή την ε, τεράστια κλίμακά τους, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και με διαφορετικό τρόπο στα ζητήματα διάσωσης, ε, βάζοντας το ερώτημα αν ε, και τα μέσα διάσωσης είναι επαρκή, αλλά και αν είναι λειτουργική η ε, θέση σε λειτουργία τους σε παρόμοιες στιγμές. Ευχαριστώ. Thank you very much. Finally, Commissioner, Κύριε Επίτροπε, να πω και εγώ τα τελικά σχόλια. Πολλοί είπαν ότι το πλοίο αυτό έπλεε πολύ κοντά στην ακτογραμμή. Ε, αυτό είναι πολύ ήπιος τρόπος να το θέσουμε. Είναι από τους πιο ήπιους τρόπους που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ε, σαΐνι για να καταλάβει ότι είναι πολύ κοντά. Το θέμα είναι τι έγινε μετά. Άκουσα κάποιους που λένε μεταξύ τους, αλλά και στο κοινό και σε εφημερίδες, ότι είναι πολύ εύκολο να συλλητεύουμε σε αυτήν την κατάσταση, να κατηγορούμε ότι αυτό στέει, ο άλλος στέει κτλ. Από τη δική μου εμπειρία, όταν ασχολήθηκα με μεταφορικές, μεταφορικά ατυχήματα και καταστροφές, ε, έχω, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι καλό είναι να περιμένουμε το αποτέλεσμα της επίσημης έρευνας, να διαβάζουμε το πόρισμα, το αναλύουμε και τότε αποφασίζουμε αν χρειαζόμαστε περισσότερη ή λιγότερη νομοθεσία, αν θα πρέπει να κλείσουμε κάποια κενά που έχει νομοθεσία ε, ή αν πρέπει να πούμε ότι απλώς πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά την ισχύουσα νομοθεσία. Φαντα... Φανταστείτε τώρα τα τα μέσα ενημέρωση, α πούμε, οι εφημερίδε κτλ. τρελαίνονται να λένε αυτό στέει, α πούμε, ειδικά από την πρώτη μέρα. Εμεί ω επιχε... επαγγελματίε των μεταφορών θα πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό και να του πούμε περιμένετε το αποτέλεσμα τη επίσημη έρευνα ε, για να δούμε μετά ε, τι θα χρειαστεί να κάνουμε. Φυσικά, στο μυαλό μα είναι τα θύματα και οι οικογένειε εκείνων που έχασαν ανθρώπου μέσα αυτή την τρομερή ε, τραγωδία και τους ανθρώπους εκείνους που επιβίωσαν από αυτή την τραυματική εμπειρία. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, ερωτήσεις σας. Όπως είπα, ε, τρέχει μία έρευνα ως ε, μέλη της Επιτροπής αυτής, είπατε και εσείς Πρόεδρε, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτή την έρευνα. Οπότε αυτό νομίζω ότι απαντά στο αν τηρήθηκαν οι κανόνες ή όχι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αμφιβολίες για το αν τηρήθηκαν οι κανόνες. Τώρα, για την ρότα του πλοίου. Η ΕΜΣΑ έδωσε αμέσως χάρτες για το, όπου δείχνει ότι, δείχνουν ότι μάλλον άλλαξε ρότα το πλοίο από την πορεία που έπρεπε να πάρει ίσως ή από αυτή που ακολουθούσε η ίδια ε, εταιρεία ε, που οργάνωνε την κρουαζιέρα. Αλλά βεβαίως αυτό είναι θέμα του καπετάνιου. Ο καπετάνιος έχει τις πληροφορίες για να αξιολογήσει ποιος είναι ο, ποια είναι η καταλληλότερη ρότα για να πάρει. Ίσως αν υπάρχει από τη μία πλευρά πολύ αέρας να πρέπει να πάει από ε, μια άλλη, ε, να κάνει μια άλλη επιλογή. Οπότε αυτό είναι θέμα που θα το, δει, θα το μελετήσει η έρευνα που κάνουν οι Ιταλικές αρχές. Βεβαίως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για τον επαγγελματισμό που δείχνουν και τη δέσμευση που δείχνουν οι Ιταλικές αρχές και Βεβαίω ε, θα έχουμε όλες τις απαραίτητε πληροφορίες από την πλευρά του. Ε, επίσης, ε, το θέμα της, των μεταφορών των θαλασσίων Πάντα βεβαίω η αρχή απαράβατη είναι ότι ο καπετάνιος φεύγει τελευταίο από το πλοίο. Δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσαμε στην νομοθεσία μας να βάλουμε μια τέτοια παράγραφο που να λέει ότι ο καπετάνιος φεύγει τελευταίος. Τι να σας πω, αυτό είναι πάλι θέμα της έρευνας. Ε, όπως επίσης και το θέμα του μαύρου κουτιού. Όλοι διαβάζουμε τα νέα, τις εφημερίδες. Και πρέπει να πω ότι ήδη σκεφτόμαστε το θέμα των εκενώσεων και των κανόνων εκένωσης, αν ήταν επαρκής ή αν θα πρέπει να κάνουμε κάποιες τοποποιήσεις αλλά η εκένωση είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα σε αυτά τα μεγάλα επιβατικά πλοία. Όχι μόνο τα κροσγερόπλια, αλλά και τα επιβατικά. Υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης το οποίο δοκιμάζεται, γίνεται ε, έλεγχος των, της κατάρτισης των ε, ναυτικών συχνά και βεβαίως πάντα η απώλεια ζωής είναι τραγωδία. Ε, σχεδόν 30 άνθρωποι έχουν χάσει την ε, ε, ζωή τους, αλλά ε, περίπου 4.000 άνθρωποι βγήκανε σώοι από το πλοίο. Μην το υποτιμούμε και αυτό. Οπότε βεβαίως τα νέα δείχνουν μόνο τον πανικό και προφανώς αν ήμασταν και εμείς σε μια τέτοια κατάσταση, ε, δεν θα ήμασταν και πολύ ψύχρεμοι, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά οι περισσότεροι βγήκανε ζωντανοί από το πλοίο με τη βοήθεια του ε, πληρώματος. Οπότε και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί θετικά. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι το θέμα δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, και αυτό βεβαίως ερευνάται. Τώρα για την κατάρτιση, για την εκπαίδευση του πληρώματο. Και αυτό βεβαίω είναι πολύ σημαντικό και όλοι φυσικά ενδιαφέρονται για την ασφάλεια σε αυτά τα μεγάλα κροσγερόπλια. Επίση, ένα ερώτημα που ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, που το ρώτησε κάποιο από εσά είναι μήπω πρέπει να μειώσουμε το μέγεθο αυτών των επιβατικών πλοίων ή ακόμη και των κρουαζιεροπλοίων. Ε, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εξ ορισμού το μέγεθο είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Αν το μέγεθο έχει τη σωστή, αν το πλοίο έχει το μέγεθο αυτό που έχει, αλλά έχει τη σωστή κατασκευή, όπω ε, και τηρεί τι προποθέσει από τη Σύμβαση Σόλα, μετά από, την, ε, ε, μετά από το Τιτανικό, μετά από, την, ε, από το δυστύχημα στην Εστονία με άλλο ένα πλοίο που βυθίστηκε, τροποποιήθηκε η σύμβαση όλα. Για, ακριβώς για να αποφευχθούν τα δυστυχήματα στο μέλλον. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το μέγεθος είναι επιχείρημα που μπορεί κανείς να πει 4.000 επιτρέπεται να μπουν, 6.000 δεν επιτρέπεται να μπουν σε ένα τέτοιο μέγεθος πλοίου. Αλλά βεβαίως πρέπει να το αναλύσουμε σοβαρά, γιατί βεβαίως ε, κοινή λογική λέει ότι είναι ένα πλοίο πολυτελεία προσφέρει κάθε είδου υπηρεσία. Ε, οπότε πώς βγαίνει κανείς από αυτό το πλοίο εάν γίνει κάτι σοβαρό αυτό είναι λογικό ερώτημα. Βεβαίως πρέπει να το σκεφτούμε, είναι πολύ σημαντικό και ως προς αυτό ενημερωνόμαστε ε, τακτικά και επίσης για τα δικαιώματα των επιβατών έχουμε την Σύμβαση της Αθήνας για τις αποζημιώσεις. Αλλά βεβαίω τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, ε, υπογράψει αυτή τη σύμβαση, αλλά υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Πρώτη του 2013 ως προς αυτό. Οπότε επιτρέπεται ε, η, αποζημίωση για, τέτοιες, για τέτοια δυστυχήματα με βάση την Ιταλική νομοθεσία. Αλλά τα κράτη-μέλη που έχουν ε, ε, κυρώσει την σύμβαση της ε, Αθήνας βεβαίως μπορούν να δώσουν την αποζημίωση. Υπάρχει ένα ποσό γύρω στα 21.000 ευρώ. Πόσα μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση αυτή. Η Ιταλία δεν την έχει επικυρώσει ακόμα. Ε, συγγνώμη, ε, απλώ αναρωτιέμαι πόσα κράτη-μέλη δεν την έχουν επικυρώσει αυτή την σύμβαση. Πολλά από τα κράτη-μέλη δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Έχουμε βεβαίω τώρα εισαγάγει ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία περιλαμβάνει τον ίδιο κανόνα και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Πρώτου του 2013 για να αποφύγουμε να περιμένουμε την ε, επικύρωση των κρατών μελών. Οπότε τα δικαιώματα των ε, επιβατών θα μπορούν να εξασκηθούν. Βεβαίω για του ανθρώπου που έχασαν του δικού του, ε, δεν του δίνει και μεγάλη παρηγοριά αυτό. Α, ο ρόλος της ΕΜΣΑ. Ε, για την κατάρτιση είναι σημαντικό. αλλά ο ρόλος της ΕΜΣΑ γενικώ και στα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντικός. Τα κράτη-μέλη συχνά αντιδρούν όταν τους λέμε ότι η ΕΜΣΑ θα αναλάβει κάποιες, ε, ε, κάποια καθήκοντα ε, περιπολιών στις εκτογραμμές τους. Υπάρχουν βεβαίως και περιβαλλοντικά θέματα, εποπτείας θέματα, η ΕΜΣΑ τα έχει καταφέρει αρκετά καλά. Επίσης η μόλυνση είναι θέμα το οποίο άπτεται των αρμοδιότητων της ΕΜΣΑ. Αλλά πρόσφατα κάναμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για τη διεύρυνση της εντολής της ΕΜΣΑ και η συζήτηση αυτή πρέπει να πω ότι ήταν ε, αρκετά έτσι σαφής, υπήρξε αρκετός ενθουσιασμός, ε, γιατί προς το παρόν η εντολή που έχει η ΕΜΣΑ είναι αρκετά περιορισμένη. Οι έρευνες γίνονται από τις, από τις ε, Ιταλικές αρχές όλα τα διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές. Όπως και για, τα, για τις περιπτώσεις της ε, αεροπλοεία και των σχετικών δυστυχημάτων. Okay, so, thank you, Commissioner. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα τη ανταλλαγής απόψεων με τον Επίτροπο Κάλλας για το αεροπορικό πακέτο. Σας δίνω λίγο χρόνο να πιείτε νεράκι και να συνεχίσουμε με το πακέτο των αερομεταφορών. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ όσοι φύγουν από την αίθουσα να το κάνουν με ήσυχο τρόπο. Δεν χρειάζεται να κάνετε πηγαδάκια για να δίνετε διαλέξεις όσο βγαίνετε από την αίθουσα. Okay. Honorable members. Αγαπητοί και αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, το αεροπορικό πακέτο Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, των αερολιμένων, ενισχύοντας το δυναμικό τους και βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Να περιμένουμε λίγο για να αδειάσει αίθουσα. <laughs> Εκένωση, εκένωση. με τα σλότς, τις χρονοθυρίδες. Το ισχυρό σύστημα για τις χρονοθυρίδες και την κατανομή τους θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό. Τα πιο κομβικά αεροδρόμια δεν ε, αξιοποιούνται κατάλληλα το ισχύον σύστημα δεν είναι αρκετά ελαστικό για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη κίνηση στα αεροδρόμια. Γι' αυτό θα πρέπει να προαγάγουμε την κινητικότητα των χρονοθυρίδων με το δευτερογενέ εμπόριο. Δηλαδή, οι, οι αεροπορικέ εταιρείε μεταξύ του θα πρέπει να μπορούν να κάνουν αγοραπολισίε χρονοθυρίδων σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο. Δευτερογενές εμπόριο, το δευτερογενέ εμπόριο θα εξασφαλίσει καλύτερη αξιοποίηση των χρονοθυρίδων μεταξύ των αεροπορικών εταιριών και θα αποσυφορήσει τα πιο κομβικά αεροδρόμια. Θεωρούμε ότι ε, και μόνο οι αλλαγές στις χρονοθυρίες επιτρέψουν την αύξηση μέχρι το 2025 των ετήσιων μεταφορών κατά 25 εκατομμύρια επιβάτες. Έχουμε Επίσης θα κοστίσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ και ε, πολλές θέσεις απασχόληση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Χρειαζόμαστε και πιο διαφανείς πληροφορίες και καλύτερες πληροφορίες για το ποιο είναι ο ιδιοκτήτης, ο κύριος των χρονοθυρίδων σε κάθε αεροδρόμιο. Άλλα στοιχεία της πρότασης ε, των χρονοθυρίδων είναι να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των συντονιστών των χρονοθυρίδων σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες εδάφους, ground handling. Πολύ συχνά ε, η ποιότητα υπηρεσιών εδάφους επηρεάζουν τις καθυστερήσεις. Χρειαζόμαστε αξιοπιστία, ακρίβεια στις πτήσεις και διαφάνεια και για το κόστος. Βέβαια έχουμε ένα δυναμικό εμβόλιο υπηρεσιών εδάφου ε, που απασχολεί πάνω από 60.000 ε, εργαζόμενους, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα των υπηρεσιών εδάφου ε, και ως προς την αποτελεσματικότητα και ως προς την ποιότητα. Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει περισσότερη επιλογή Απελευθέρωση λοιπόν θέλουμε των υπηρεσιών εδάφους και να έχουμε τουλάχιστον τρεις παρόχους υπηρεσιών σε κάθε αεροδρόμιο. Δηλαδή πάνω από 5 εκατομμύρια ε, επιβάτες το χρόνο, γιατί από ένα τέτοιο μέτρο θα υποφεληθούν κυρίω οι επιβάτε. Επίση, οι αεροπορικέ εταιρείε θα πρέπει να, κάνουν μόνες, να μπορούν να αναλάβουν μόνε του τι ε, υπηρεσίε εδάφου, το self-handling δηλαδή, κάτι που δεν ισχύει σε όλα τα αεροδρόμια σήμερα. Θέλουμε και καλύτερο συντονισμό του ground handling των υπηρεσιών εδάφου στα αεροδρόμια. Και πιστεύουμε ότι καλύτερα αρμόδια για αυτό το συντονισμό είναι τα αεροδρόμια τα ίδια. Βέβαια, δεν θα πρέπει ο ανταγωνισμό να οδηγήσει σε μια υποβάθμιση τη ποιότητα. Θέλουμε κάποια ποιοτικά κριτήρια προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη των προδιαγραφών. Τελευταίο θέμα για το ground handling αφορά το προσωπικό εδάφους. Οι ποιοτικέ υπηρεσίε προποθέτουν φυσικά καλού επαγγελματίε. Δηλαδή, θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε του όρου ε, Σταθερό ηθικών εργασία για το προσωπικό εδάφους. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τις απαιτήσει για την πρόσληψη προσωπικού εδάφους και να υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις για ελάχιστη εκπαίδευση ή κατάρτιση του προσωπικού εδάφους. Τέλος, για την χορύπανση. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, συμπολίτες μας από υπερβολική χορύπανση, ιδιαίτερα όσους κατοικούν κοντά σε αεροδρόμια. Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι οι αποφάσεις για τη μείωση του επίπεδου θορύβου θα πρέπει να είναι ισορροπημένες. Γιατί έχουμε αφενός την προστασία των ε, κατοίκων που βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια και αφετέρου το συμφέροντα των επιβατών αυτή η ισορροπία θα πρέπει να διέπει την επιλογή των ε, κατοφυλίων ήχου. Έτσι και οι αρμόδιες αρχές ε, θα πρέπει ε, να καταλήξουν ρυθμίσεις για να αποφευθεί υπερβολικό επίπεδο θορύβου. Αυτό είναι το πακέτο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο ε, ωραίο, μια τέτοια ωραία νομοθετική πράξη και τελικά την, ε, ε, την πράξη αυτή θα την ψηφίσει μόνο η Κομισιόν. Ε, ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Κομισιόν και ε, Κοινοβουλίου. Ο Επίτροπος πρέπει να φύγει σε λίγο, αλλά θα μείνει όσο μπορεί περισσότερο. Θα τραβήξουμε λίγο την παραμονή του. Ο κύριος Λάιτφριντ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε είχαμε αμφιβολίες. Είχαμε αμφιβολίες για το αν αυτό το πακέτο θα μπορέσει να κάνει πιο ελκυστικές τις πτήσεις και τα αεροδρόμια. Οι αμφιβολίες μας αυξήθηκαν. Ε, μιλούμε για τη ρύθμιση των χρονοθερίδων. Εντάξει, θα τη συζητήσουμε στο, στην λεπτομέρεια του, αλλά θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Γκρό. Έχει νόημα όλο αυτό. Για το θόρυβο τώρα, την ηχορύπανση. Εγώ ήμουν εισηγητή και υπάρχουν και εκεί κάποια θέματα που πρέπει να λυθούν. Όπως γιατί περιοριζόμαστε, περιορίζεστε μάλλον στην πρόταση της Κομισιόν στην καταγραφή των μέτρων. Γιατί δεν σκέφτεστε να θέσετε και κάποιους στόχους. Δηλαδή νομίζω ότι το ένα ε, ε, ε, το, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άλλο. Έχουμε πολύ σωστή, έχουμε συγκέντρωση, μάλλον πολύ αυστηρή συγκέντρωση των μέτρων στην ε, Κομισιόν για την περιορισμό του, α, ε, της συγχωρήπανσης, αλλά δεν έχουμε στόχο. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει ένας στόχος για να επιτευχθεί. Επίσης, υπάρχει, ε, υπάρχουν πάρα πολλές κατοξιδότητες πράξεις για την ψήφιση όλων αυτών και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμα όλα αυτά. Δηλαδή το κοινοβούλιο θα μείνει απ' έξω από όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες παρέμβασής μας. Και επίσης, οι υπηρεσίε εδάφους. Η ομάδα μου, αρκετοί συνάδελφοι στην ομάδα μου, έχουν πολύ σοβαρές αμφιβολίε για το κατά πόσο είναι σκόπιμη αυτή η πρόταση, στο σύνολό της. Μέσω τη πρόταση αυτή κατά τη δική μου άποψη, δεν υπάρχει καθόλου βελτίωση τη ποιότητα. Υπάρχει μάλιστα υποβάθμιση τη ποιότητα. Οι δουλειέ ε, πληρώνονται με πολύ μικρότερου μισθούς, οι υπηρεσίε είναι χειρότερε. ο καθένας θα προσπαθήσει να βρει ίσως και μια δεύτερη δουλειά για να μπορέσει να ζήσει. Αυτό γίνεται πάντα όταν στα αεροδρόμια υπάρχει απελευθέρωση των ε, υπηρεσιών ε, εδάφους. Δεν καταλαβαίνω. Εφόσον ξέρετε πώς έχει λειτουργήσει το σύστημα μέχρι τώρα, που δεν έχει λειτουργήσει σωστά, γιατί κάνετε τέτοια πρόταση. Αν θέλετε να βελτιώσουμε την ποιότητα. Το μόνο που κάνει αυτή η πρόταση είναι να μπορέσουν κάποιοι να εισπράξουν περισσότερα χρήματα και να μπουν στην αγορά ω εταιρείε, ω επιχειρήσει. Αλλά δεν βοηθάει αυτό ούτε τον επιβάτη, ούτε βελτιώνει τι υπηρεσίες που λαμβάνουν οι επιβάτε και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ξεφεύγεται από αυτό το σκεπτικό. Η κυρία Μάισνερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει η Κομισιόν, ότι θέλουμε έναν ενιαίο αέριο χώρο, το έχουμε πει και εμείς, όλα τα κρατημέλη και το θέμα είναι πώς μπορούμε παράλληλα με αυτόν τον ενιαίο αέριο χώρο να ρυθμίσουμε και τις ε, ε, δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα. Θα υπάρξει περισσότερη βεβαίως ε, διακίνηση αεροπορικών, επιβατών αεροπορικός, οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα τρία αυτά πακέτα. Μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους που θέλουμε με αυτό που προτείνουν τα πακέτα. τα, οι χρονοθυρίδες είναι αυτό που μου προκαλεί τα λιγότερα προβλήματα και αμφιβολίες τελικά παρόλο που υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες από εμπλεκόμενους φορείς, αλλά Γι' αυτό θα σας μιλήσει και ο εισηγητής μας. Το, οι υπηρεσίε εδάφους ε, με τα χρονοθυρίδες, ε, εντάξει, ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό. Τώρα, για τις ε, υπηρεσίε εδάφους. Είναι κρίμα που γίνεται τόσο θερμή η συζήτηση, προφανώς δεν θέλουμε να, να πληγεί η ασφάλεια. Προφανώς θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο με αυτή την, με αυτή την πρόταση. Και 70% των καθυστερήσεων των πτήσεων γίνεται λόγω των καθυστερήσεων στις υπηρεσίες εδάφους. Οπότε, με τις προτάσεις αυτές που κάνουμε μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, δηλαδή να έχουμε λιγότερες ε, καθυστερήσεις. Εν τω μεταξύ έχει υπάρξει και άλλη μια έκθεση από τη δική μας την ομάδα, από την Επιτροπή ε, Μεταφορών και είδαμε ότι σε κάποιους τομείς γίνεται δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Σε άλλου τομεί πάλι μπορούμε να μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί εδώ προτείνεται κανονισμός ο οποίο είναι άκαμπτο ε, εργαλείο. Μια οδηγία είναι λίγο πιο ευέλικτη. Μπορεί να περιλάβει πολύ περισσότερα στοιχεία και να προσαρμοστεί πολύ καλύτερα στι ε, ιδιαιτερότητε του κάθε αεροδρομίου. Επίση, καλό είναι που μιλάτε για τα κριτήρια ποιότητα, τα οποία είναι σκόπιμα, είναι λογικά και βεβαίω ε, θεωρώ ότι θα μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Θα μπορούσαν. Για τον χορύπανση τώρα. Ε, εμείς ε, έχουμε πραγματικά κατακεραυνοθεί από email που λαμβάνουμε, σημειώματα, ε, εμείς οι Γερμανοί εννοώ, ε, διαβάζουμε συνέχεια άρθρα, δίνεται η εντύπωση, και κλείνω πρόεδρε, ότι η οικονομία είναι πάνω απ' όλα και οι, η των κατοίκων που ζουν κοντά σε περιοχές με αεροδρόμια δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε λοιπόν εδώ μια ισορροπία. Ε, αυτό με, που αποφασίζουμε τελικά θα λύσει το πρόβλημα γιατί προφανώς θέλουμε ας πούμε στην ε, Φραγκφούρτη υπάρχει ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Αν επιβαρυνθεί ή αν περιοριστεί πολύ περισσότερο το αεροδρόμιο της ε, Φραγκφούρτης, προφανώς θα πληγούν ε, άνθρωποι, θέσεις εργασίας κτλ. Απ' την άλλη όμως δεν μπορούμε να αμελούμε και το πρόβλημα που υπάρχει με την χορύπανση στο, ε, στη Φραγκφούρτη. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Να πω καταρχάς κάτι γενικό. Πάρα πολλές κατοξιδότηση πράξεις. Δεν συμφωνώ. Αυτό το νέο εργαλείο θα το χρησιμοποιήσουμε, ε, χρησιμοποιείται μάλλον τόσες πολλές ε, κατεξιότητες πράξη για να, πως, για να ε, κλέψετε αρμοδιότητες από το Κοινοβούλιο. Διαφωνώ κάθετα. Δεύτερον, χρονοθυρίδες. Δύο μεγάλα προβλήματα βλέπω εδώ στο θέμα των χρονοθυριδών. Ε, το θέμα των δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα υπάρξει εγκαθίδρυση μονοπωλίων εκεί και τα προβλήματα θα οξυνθούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα οι, οι χρονοθυρίδες να ορίζονται ανάλογα και με την απόδοση την περιβαλλοντική. Για παράδειγμα, να δούμε την, ε, τον θόρυβο, την εκπομπή αερίων. Αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, έτσι ώστε να ε, δίνονται τα σλότς χρονοθυρίδες στα διάφορα αεροδρόμια. Επίσης, τα ψηλότερα ε, πρότυπα. Δεν έρχονται μέσω της, ε, ε, του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας μόνο, αλλά μέσω των καλύτερων, της καλύτερης επικοινωνίας. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν καλύτερη συνδεσιμότητα. Δεν μπορεί κάποιο να έχει ένα πρόβλημα και στι υπηρεσίε ελάφου, α πούμε, και κανένα να μην είναι υπεύθυνο, γιατί αυτό έχει επιπτώσει και στον επιβάτη. Τώρα, για τις αρμοδιότητες, για τα ενασφάλεια και το περιβάλλον. Όσο περισσότερα διαχωρίζουμε τα, τους τομείς, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρει κανείς, την, να βρει κανείς υπεύθυνο. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς στην Γερμανία οργανωμένη ανευθυνότητα. Ιδιαίτερα προβληματικό θεωρώ ότι είναι αυτό το σκεπτικό που υπάρχει για την ηχορύπανση εδώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα ιδιαίτερα, τα τοπικά χαρακτηριστικά, όχι μόνο για το θόρυβο. Αυτό είναι προφανώς πολύ σημαντικό. Και αυτό θα πλήξει τους α, πολίτες που ζουν στα, κοντά στα αεροδρόμια. Πρέπει να ληφθούν λοιπόν πιο αυστηρά κριτήρια και μέτρα αλλά πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένοι έλεγχοι και για τα, για τα health kits και επίσης ε, τέτοια, σε τέτοια θέματα πρέπει να δούμε πώς θα, το, θα τα ρυθμίσουμε. Υπάρχει η χορύπανση που σε πολλές πόλεις δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η Βιέννη ας πούμε έχει τεράστιο πρόβλημα το Ινσπρουκ επίση ε, λόγω γεωγραφική θέση έχει πολύ σημαντικά προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πακέτο θα πρέπει να είναι συνεκτικό, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με, το, με τις ε, υπηρεσίες ε, εδάφους. Αν πρέπει όντως να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα. Γιατί φαίνεται ότι σε κάποια, από κάποια στιγμή και έπειτα η απελευθέρωση δεν προσφέρει τίποτα ούτε στους πελάτες ούτε στους επιβάτες παρά μόνο προβλήματα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Όχι να κοιτάμε μόνο τα οικονομικά συμφόροντα των μεγάλων αεροδρομίων. Ευχαριστώ. Τρία λεφτά για την κυρία Φώστερ το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να μιλήσω για τις ε, υπηρεσίες εδάφους από την πλευρά τη σκοπιά του Ηνωμένου Βασιλείου, εμείς πάντα εφαρμόζαμε χαλαρούς κανόνες στις εταιρείε για τους, τις υπηρεσίες εδάφους. Για μας δεν είναι πρόβλημα. Για τους επιβάτες τώρα έχουμε ανησυχίες. Ε, ορισμένοι, ορισμένες εταιρείε χρησιμοποιούν το προσωπικό που έχει το αεροδρόμιο, άλλε εταιρείε χρησιμοποιούν το δικό του προσωπικό και επομένω ο επιβάτη δεν ξέρει ποιο έχει την ευθύνη. Υπάρχουν συγκρούσει ανάμεσα στι εταιρείε και στο αεροδρόμιο τελικά. Πρέπει να έχουν σωστέ πληροφορίε οι επιβάτε, νομίζω. Επίση, ε, σταθερή α, δουλειά για το προσωπικό, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, για το θέμα των χρονοθυρίδων. Για μας το μεγαλύτερο, για το, μεγαλύτερο είναι το Heathrow. Συχνά ε, πολλά εξαρτώνται για, το πώς λειτουργεί δηλαδή το αεροδρόμιο από το πώς κατανέμουν τις χρονοθυρίδες οι υπεύθυνοι συντονιστές. Ε, πρέπει να είναι σίγουρο ότι παίρνουν σωστές αποφάσεις. Ε, επίσης, πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες ή όχι, απλώς να τους εφαρμόσουμε σωστά. Έπειτα, ε, υπάρχουν και τρίτες χώρες που επηρεάζουν το τι συμβαίνει στην ε, Ευρώπη. Τώρα, όλοι εφαρμόζουν τον 80-20. Ε, Το βασικό είναι να χρησιμοποιούν σωστά οι εταιρείε τα... τις του. τους. Όταν έχουμε ας πούμε, προβλήματα με την ηφαιστειακή ε, σκόνη, α, υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με την κατανομή των χρονοθυρίδων. Άλλο είναι να έχει μια χρονοθυρίδα μία στις 20 και άλλο μία στις 5 για τον κανονισμό ε, για την ηχορύπανση. Ε, δεν ξέρω, υπήρχε παλιά οδηγία και τώρα έγινε καονισμό. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει ένα θέμα όμως επικουρικότητα εδώ. Ε, νομίζω ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συναποφασίζουν για το ότι είναι σημαντικό για τα δικά τους ε, αεροδρόμια. Επίσης για τη χρήση της γης. Ε, είναι τεράστιο θέμα ε, με το το πού θα χτιστούν τα αεροδρόμια, ή αεροδρόμια τα οποία υπήρχαν ήδη, επίσης για το πώς θα μειωθεί ο θόρυβος, τα μέτρα αυτά για τη μείωση του θορύβου. Έχουμε μέτρα όπως το ΣΕΖΑΡ που, που λειτουργούν. Για το κεφάλαιο 3, κεφάλαιο 4 για τα αεροπλάνα. Δεν θα ήθελα αεροπλάνα όπως τα Α320 να παροπληστούν, ας πούμε, γιατί των κάποιος θα θεωρήσει ότι δεν πληρούν όλους τους κανόνες. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα των αεροπλάνων που οριακά ε, δεν πληρούν τους κανόνες. Ε, τελειώνω τον πρώτο γύρο με τον κύριο Κόχλιτσεκ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε τις τρεις οδηγίες η Ευρώπη δεν θα πρέπει να απομονωθεί από τις υπόλοιπε χώρε του κόσμου. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. υπάρχει θέμα συντονισμού. Επίσης και στον τομέα του θορύβου και στον τομέα της ε, κατανομής των, των ε, αυτό επηρεάζει τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα. Το τρίτο θέμα, οι υπηρεσίε εδάφου. Υπάρχει θέμα κόστους και θέμα μέσων. Επίσης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί Πρέπει να δούμε τι απελευθέρωση επιτρέπουμε, τι χαλάρωση των κανόνων επιτρέπουμε. Επίση, θα πρέπει οι κοινωνικέ συνθήκε εργασία των εργαζομένων να είναι σωστέ, να υπάρχει ένα ορισμός για αυτές και θα πρέπει όλο το προσωπικό να έχει τη σωστή κατάρτιση. Θα πρέπει να έχουμε τέτοιου κανόνε, γιατί αλλιώ θα χαθούμε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ανταγωνισμό. ε. Θα διαβάσατε ότι το 30% της, ε, των αεροπορικών ροών είναι στα χέρια της Ευρώπης. Το υπόλοιπο 70% είναι στα χέρια των ξένων. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε στο πρώτο γύρο, γιατί ξέρω ότι μετά πρέπει οπωσδήποτε να φύγετε. Αλλά φύγετε στο πόδι σας τον κύριο Μπάλντουιν. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να οριστικοποιήσουμε αυτή την πρόταση και να καταλήξουμε σε νομοθετικές ε, διατάξεις. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και στο μέλλον να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Αφήνω πάντως ε, στο πόστο μου τον κύριο Μπόλτουιν που είναι διευθυντής για θέματα αεροπλοείας. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω τα τρία βασικά ζητήματα που επισημάθηκαν στη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων. Το θέμα των χρονοθύριδων καταρχήν, των σλότς. Εγώ αρχικά δεν ήξερα τι είναι χρονοθυρίδα και τι σημαίνει διάταξη ή ρύθμιση για χρονοθυρίδες. Εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν μια αεροπορική εταιρεία αγοράζει ή κάνει σύμβαση με το αεροδρόμιο για απογείωση, προσγείωση και χρήση ε, των υπηρεσιών, αυτό ε, συμπεριλαμβάνεται στο σλότ. Το σλότ όμως είναι μόνο δικαιώματα απογείωσης προσγείωσης και τα διαχειρίζεται ένας συντονιστής. Ε, δεν έχει καμία σχέση με την αγορά, μια ειδική συντονιστική ρυθμιστική αρχή. Βέβαια, όταν το αεροδρόμιο δεν είναι υπερβολικά γεμάτο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως ε, υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία, τότε είναι πολύ πιο δύσκολη η κατανομή των χρονοθυρίδων. <clears throat> Και σε μερικές περιπτώσεις έχουμε πολλά τεχνητά εμπόδια ε, που αναχαιτίζουν την καλύτερη χρήση των δικαιωμάτων ε, απογείωσης προσγείωσης και των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή των σλότ ουσιαστικά. Έχουμε καταθέσει δύο προτάσεις για συζήτηση. Η μία αφορούσε τον πληστηριασμό. Αρχικά είχαμε προτείνει να καταργήσουμε όλους τους μηχανισμούς για τις χρονοθυρίδες και να ξεκινήσουμε τα μπουλεράζα του μηδενός με δημοπρασία. Βέβαια αυτή η πρόταση παραθεωρήθηκε, θεωρήθηκε υπερβολικά μεγάλη επίβολη και είπαμε εντάξει, δημοκρασία, δημοκρασία μόνο για τις νέε χρονοθύριδε, όταν υπάρχει διεύρυνση του δυναμικού. Αυτή ήταν μια άλλη εναλλακτική λύση. Αλλά και εκεί προσκρούσαμε σε αντιστάσεις, σε δρυμύτατε κριτικέ από όλους τους ενδιαφερόμενους. για ευνόητους λόγους, γιατί θα ήταν δύσκολο να προσδιορίσουμε το νέο δυναμικό, τη νέα ικανότητα, το θέμα της χρηματοδότησης. Οπότε εγκαταλείψαμε και αυτή την πρόταση και καταλήξαμε στην πρόταση για το secondary trading, το δευτερογενές εμπόριο, δηλαδή να μπορούν οι αεροπορικές εταιρείε μεταξύ τους να τα διαπραγματεύονται τα σλότ. Και συμφώνησαν και οι αεροπορικέ εταιρείε και τα αεροδρόμια. Πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση θα λειτουργήσει εύρυθμα. Οπότε μία αεροπορική εταιρεία δεν θα χρειάζεται να κρατάει τα σλότ για τους λόγους της, επειδή τους χρειάζεται στο μέλλον ε, θα τις χρειάζεται στο μέλλον τις χρονοθυρίδες. ή θα συντηρεί γατρικές μόνο και μόνο για να κατακρατούν χρονοθυρίδες. Ήταν λοιπόν πολύ θετική η αντίδραση. Τώρα, το 85-15 είναι προσυζήτηση για το ποιο θα είναι το τμήμα αυτού του δεύτερου γενούς εμπορίου. Δεύτερο ζήτημα, η υπηρεσία σε δάφος, το ground handling. Όπω σας είπα, υποβάλαμε και τις σχετική ανακοίνωση και διαπιστώσαμε ότι τρει στι τέσσερι καθυστερήσει ε, πτήσεων οφείλονται σε προβληματικέ ε, υπηρεσίε εδάφου. Γι' αυτό θέλουμε αναβάθμιση τη ποιότητα ε, των υπηρεσιών εδάφου για να περιορίσουμε και τι καθυστερήσει. Άλλωστε υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ των αεροδρομίων, υπάρχει διαφορετική οργάνωση. <clears throat> Είναι πολύ μορφό το τοπίο στα αεροδρόμια και όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα Βελτίωση των υπηρεσιών εδάφους προκειμένου να περιοριστούν και καθυστερήσεις. Τρία είναι τα πιο βασικά στοιχεία στη συζήτηση και στην πρόταση. Καταρχήν υπάρχουν ε, απαιτήσεις για προδιαγραφές ποιότητας. Πολύ το επισημάνατε και συμφωνώ και εγώ ότι δεν θα πρέπει να γίνει μία εξίσωση προς τα κάτω. Δεν είναι θέμα κόστος μόνο, υπάρχει και θέμα ποιότητας δεν θα πρέπει να γίνει υποβάθμιση. Επίση, δεν θα πρέπει επιβάτη να χάνει την αποσκευή του. Όλε αυτέ οι προδιαγραφέ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ποιότητα. Θα δούμε πώς θα τις ε, διατυπώσουμε. Υπάρχει και το κοινωνικό ζήτημα των δικαιωμάτων των ε, παρόχων υπηρεσιών εδάφους. Είχαμε εκτενέστατες συζητήσεις με την ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές και μας είπε η Ομοσπονδία αυτή ότι αν έχουμε περισσότερη ελαστικότητα και περισσότερες εταιρείε, θα έχουμε πολύ πιο εύκολες απολύσεις. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλεψη στην πρότασή μας. Ένα είδος κοινωνικής πρόβλεψης, κοινωνικής διάταξης, για να αποφευθούν τέτοιες ε, εύκολες απολύσεις και θεσπίζονται κάποιοι κανόνες προκειμένου να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος και η πιθανότητα τέτοιων αλλαγών. Δεύτερο στοιχείο του πακέτου για τις υπηρεσίες εδάφους είναι ότι εμείς προτείνουμε μόνο στα μεγάλα δρόμια αύξηση των παρόχων υπηρεσιών από 2 σε 3 και μπορώ να σας κατονομάσω ποια αεροδρόμια αντιτάχθηκα στην πρόταση αυτή είναι σίγουρα λιγότερα από δέκα τα αεροδρόμια που εξέφρασαν αστάσεις και γνωρίζω θαυμάσια τους λόγους για τους οποίους διαφώνησα τα αεροδρόμια. Και ήδη επισήμαναν το πρόβλημα και στους υπουργού. Αντιτάχθηκαν τα αεροδρόμια γιατί λύνουν και δένουν, ελέγχουν πλήρως τις υπηρεσίες εδάφους. Αν όμω πει κάποιο ότι αυτό είναι καλό για τι υπηρεσίε και καλό για την ποιότητα, δεν το θεωρώ ότι αυτό το μονοπόλιο είναι καλό, εκ μέρου ορισμένων αεροδρομίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα θορύβου, την ηχορύπανση, καλύψατε όλα τα στοιχεία, όλε τι πτυχέ τη ηχορύπανση. Σίγουρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο θόρυβος είναι ένα στοιχείο της ρήπανσης που θα πρέπει να περιοριστεί, να καταπολεμηθεί, να προσδιορίσουμε κάποιες προδιαγραφές για να περιορίσουμε το θόρυβο και την ηχορύπανση. Υπάρχουν όμως και κάποιες τεχνικές διατάξεις. Οι κατασκευαστές ε, και αεροναυπηγοί λαμβάνουν υπόψη αυτό το θέμα και στο Μπουρζέ είχαμε μια απογείωση Α380 και κρίθηκε ε, ποια είναι η διαφορά στα επίπεδα θορύβου μεταξύ απογείωση στρατιωτικού αεροσκάφους και απογειωση ε, α Α380 ήταν πολύ φυσικά μεγαλύτερη χορύπαση από τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Θα πρέπει πάντως να περιορίσουμε την ηχορύπανση αλλά ταυτόχρονα να μην στρεβλώσουμε την εύρυθμη λειτουργία ε, του αεροδρομίου. Δηλαδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε κλείους ασφαλείας γύρω από το αεροδρόμιο παρακολύοντας την ε, σωστή λειτουργία του. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των ε, κατοίκων της περιοχής αλλά και των συμφερόντων των αεροδρομίων. Έχουμε και θέματα ανταγωνισμού, όπως είπε ο κ. και Δεν μπορούμε να είμαστε ε, υπερβολικά φιλόδοξοι. Έχουμε κάποια αεροδρόμια ε, στη Μέση Ανατολή που εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο και δεν θέλουν κουβέντα για επίπεδα θορύβου. Έχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε με τους ομιλητές γιατί θα μας αφήσει ο Επίτροπος. Παρακαλώ να περιοριστείτε στο δίλεπτο όλοι. Ξεκινώ από την κυρία Ντεβεϊράκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο Ματιό Εγκρός, η πιο απλή λύση θα ήταν να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη νέων υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έτσι δεν θα χρειαζόταν να ανασκουμποθούμε και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των, της βελτιστοποίησης ε, των, υπαρχουσών ε, υποδομών. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Θα ήθελα να πω ε, δύο λόγια για τις τρεις πτυχές του πακέτου, για την βοήθεια στη σκάλα. Ε, η αναθεώρηση έχει φέρει καρπούς. Ε, ε, είναι και η ώρα για να επωφεληθούμε περισσότερο. έγιναν σοβαρές προσπάθειες από τα αεροδρόμια τα τελευταία δέκα χρόνια για να ανοίξουν στην στην απελευθέρωση και η πρόταση της Κομισιόν είναι ισορροπημένη γενικά και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων. Για την ηχορύπανση. Πηγαίνουμε μάλλον προς σωστή κατεύθυνση από ό,τι φαίνεται, αλλά να υπενθυμίσω στην Κομισιόν ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να διατηρήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητες ε, των αεροδρομίων μας και ακριβώς γι' αυτό ε, νομίζω ότι τα κράτη-μέλη και οι τοπικές αρχές είναι οι, α, καταλληλότεροι ε, γιατί γνωρίζουν τα συμφέροντα και των επιχειρήσεων και των αεροδρομίων και θέλω να το λάβει υπόψη η Κομισιόν. Τώρα για τι χρονοθυρίδε, όπω και οι περισσότεροι συνάδελφοι, έχω κάποιε δυσκολίε. Ε, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ο στόχο που επιδιώκει η Κομισιόν. Ε, ξέρουμε όλοι μας ότι πρέπει να, αποδείξουμε, να δείξουμε ευελιξία προ τι προς τις ε, αερομεταφορές ε, σε αυτήν την περίοδο κρίση και θα πρέπει να τηρήσουμε τι δεσμεύσει μα. Όπω είπα και στα πλαίσια της ε, συμπερίληψης των αέριων μεταφορών ε, στο σύστημα ανταλλαγής ε, εκπομπών. Δεν θα πρέπει να βαρύνουμε ε, τις αεροπορικές μεταφορές με υπερβολικούς κανόνες. Θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναπνεύσουν και να περάσουν αυτή την κρίση. Για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και για την για τους κανόνες που έχουμε για τις ονοδηθυρίδες, νομίζω ότι έχουμε υπερβολικούς κανόνες πέρα από αυτούς που μπορούν να αντέξουν οι εταιρείε μας. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, δύο λεπτά. Κρίμα που έφυγε ο Επίτροπος, γιατί η ερώτησή μου ήταν απευθείας για τον Επίτροπο. Είπε να προσπαθήσει για μια μέρα έστω να μπει στη θέση ενός υπεύθυνου αεροδρομίου γιατί βρίσκονται πρωτοτελεσμένα γεγονότων πολλέ φορέ υπεύθυνοι αεροδρομίου. Οι αποφάσει λαμβάνονται ερήμην του. Τα τρία στοιχεία του πακέτου για του αερολιμένε χαρακτηρίζονται από το πρόβλημα αυτό. Και το θέμα του δυναμικού δεν είναι μόνο θέμα αγοραπολισία χρονοθυρίδων. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Υπάρχει πρόβλημα υποδομών και εκεί είναι το ζήτημα. Και δεδομένη κατάσταση των υποδομών, και σε σχέση με τις τεράστιες επενδύσεις που κάνουν οι ΗΠΑ σε αντίθεση με εμά, πώς ε, πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση στις υποδομές δεδομένης και της αντίδρασης ε, των επιβατών και των προβλημάτων της συγχωρήπανσης. Επίσης, αν έχουμε ε, σημαντικά, σημαντικούς κόμβους και κλάστερς και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Τα περιφερειακά αεροδρόμια αποτελούν το αντικείμενο γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, αλλά θα πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη ότι αφορά τη δυνατότητα διαχείριση και διοίκηση των υπευθύνων των αεροδρομίων, να, να μπορούν να ρυθμίζουν τα του οίκου του, τα του αεροδρομίου του ε, και να συμπεριλαμβάνονται στι διαβουλεύσει σε όλε τι φάσει του πακέτου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι προδιαγραφέ ποιότητα. Γιατί, επαναλαμβάνω, λαμβάνονται αποφάσει για το δυναμικό και τη χωρητικότητα των αεροδρομίων και για τις υπηρεσίες εδάφους χωρίς να ε, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι πραγματικές ε, δυνατότητες που έχει ένα αεροδρόμιο να εξέλθει από την κρίση και να κάνει καλύτερη διαχείριση της κατάστασης ή τα θέματα εχμής, ορών ε, εχμής ή ορών μικρότερης κυκλοφορίας. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Πώς λοιπόν θα εξασφαλίσει η σημαντική συμμετοχή υπευθύνων των αεροδρομίων στις ε, διαβουλεύσεις για το πακέτο, γιατί ούτως ή άλλως ε, με όποια ε, εταιρεία και να ταξιδεύουν οι επιβάτες θα χρειαστεί να περάσουν από το αεροδρόμιο του Μπαράχας, από το αεροδρόμιο των Βρυξελών και ούτω καθεξής. Ουτζίας, δύο λεφτά. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση πριν πω στην ουσία τη πρόταση. Η πρόταση τη Κομισιόν είναι καλή αφετηρία. Και για τα τρία στοιχεία του πακέτου. Αλλά όμως μπαίνουν κάποια ερωτήματα. Καταρχάς για τις χρονοθυρίδες. Η αύξηση των χρονοθυρίδων αυξάνει τον ανταγωνισμό και τη δουλειά που έχουν οι εταιρείε. Η πρόθεση της Κομισιόν είναι να δημιουργήσει φαντάζομαι μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Ε, όμως ως εργαλείο δεν είμαι σίγουρος ότι φέρνει κατά ανάγκη αυτό ως αποτέλεσμα. Έχουν γίνει κάποιες προ, για να δείτε πώς θα γίνει, θα εξασφαλιστεί αυτός ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός και μπορεί η Κομισιόν να μας δώσει αυτές τις προσωμιώσεις αν έχουν γίνει. Δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι πάτε να δημιουργήσετε μια ε, μονοπωλιακή κατάσταση των μεγαλύτερων εταιριών, διευρύνοντας τον αριθμό των πτήσεων στο εσωτερικό του, του πακέτου με, μεγαλύτερη συχνότητα δεν νομίζετε ότι τιμωρείτε τις μικρότερες εταιρείες. Άλλη ερώτηση. Πώς θα γίνει στην πραγματικότητα η ανακατονομή των ε, χρονοθυρίδων ε, σε περίπτωση που δεν έχουν σεβαστεί αυτό το 85% των πτήσεων. Δηλαδή, όταν ε, τις τιμωρείτε στην περίπτωση που δεν έχουν ε, σεβαστεί αυτό τον το 85% και γίνεται ανακατανομή των χρονοθυρίδων. Πώς ανακατανέμονται στην πράξη. Ευχαριστώ. Μάικλ Κράμερ, δύο λεπτά. Ε. ε τώρα βλέπουμε τους, ότι Σπήραμε τόσα χρόνια, Πρόεδρε, οπότε μη σας ε, εκπλήσει γιατί δεν αρκεί η δυνατότητα. Και γιατί υποστηρίζουμε τόσο πολύ την αερο, τις αερομεταφορές και μετά ε, παραπονιόμαστε για τις συνέπειες. Για την πρόταση της Κομισιόν, πάλι για λεφτά πρόκειται το κόστο είναι αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ε, ρόλο. Κάναμε την ίδια συζήτηση στη Φραγκφούρτη, ε, ε, στο Βερολίνο. Οι, οι αεροπορικέ εταιρείε αρνούνται να κάνουν μια παράκαμψη 2-3 χιλιόμετρων και να πάνε μέσω ενός άλλου μέσω ενό άλλου περιφερειακού αεροδρομίου και προτιμούν να χτιστεί ένα νέο αεροδρόμιο το οποίο θα επιβαρύνει επίση χιλιάδε ανθρώπου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πλήττονται από, την, από τις αερομεταφορές ε, και κάθε χρόνο εμείς ε, επιδοτούμε τις αερομεταφορές με 30 δις. Ε, γιατί δεν υπάρχουν λοιπόν ελάχιστα πρότυπα για κάθε, για κάθε αεροδρόμιο για την ηχορύπανση και τα οποία να πρέπει να πληρούνται. Ας πούμε, αν η Φραγκφούρτη αποφασίσει να απαγορεύσει τις νυχτερινές ε, πτήσεις, η Κομισιόν τι θα κάνει θα πρέπει να παρέμβει, δεν θα μπορεί όμω. Υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των, πιο, των, των αεροδρομίων με το μεγαλύτερη χορύπανση τελικά. Υπήρξε κάποια στιγμή στο Ζάρμπρουκεν μια ανοιχτερινή απαγόρευση. Το Ζάρμπρουκεν είπε δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε κανένα, α, κανένα αεροπλάνο να πετάξει και τελικά το κόστος το πλήρωσαν οι πολίτες της περιοχής. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ πιο προσεκτικά τα πράγματα αυτά. Τώρα οι υπηρεσίε εδάφου. Τελευταίο σημείο. Στο γερμανικό, στη γερμανική ε, Άνω Βουλή ποτέ δεν υπήρξε περίπτωση όπου όλες οι ε, πολιτικές ομάδες και, το, και οι φιλελεύθεροι ε, μαζί με, τους, ε, με τα συνδικάτα να είναι αντίθετοι με τις υπηρεσίες εδάφους. Πρωτοφανές αυτό που έγινε, οπότε δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Uh, Ähm, Ευχαριστώ. Αυτή η νέα πρόταση για τις υπηρεσίες εδάφους νομίζω ότι ε, πάει μόνο προς το συμφέρον των αεροπορικών εταιριών. Αυτοί έχουν ε, μόνο συμφέρον από αυτές τις υπηρεσίες και δεν βλέπω καμία ισορροπία μεταξύ οικονομίας και απασχολούμενων. Η πρόταση δεν φέρνει καθόλου καλύτερη ποιότητα ούτε αποτελεσματικότητα στις ε, υπηρεσίες εδάφους αν υπάρχει δηλαδή μια ακόμα ε, εταιρεία, αν ενταχθεί άλλη μια εταιρεία. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που, κάνουν αυτές, που προσφέρουν αυτέ τι υπηρεσίε να πληρώνονται καλά και να είναι εξειδικευμένοι. Έχουμε έρθει σε επαφή με τα συνδικάτα και από την Αυστρία και από τη Γερμανία και στις συζητήσεις αυτές κατέστη ε, σαφές ότι τώρα μιλούμε για 7 ευρώ την ώρα στη Γερμανία για τους ε, συναδέλφους που εργάζονται στην, ε, στις υπηρεσίες εδάφους. Αν κάποιος πρέπει να κάνει και άλλη μια δεύτερη δουλειά για να μπορεί να ζήσει, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να οξυνθεί κι άλλο. νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να έχει πολύ περισσότερο ανταγωνισμό για τις υπηρεσίες εδάφους. Ε, εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση στην, ε, στο Ανόβερο, όπου ε, τα συμβούλια μεταφορών και οι συνδικαλιστές ε, κάθισαν μαζί, συζήτησαν και όλες οι, προσωπούνταν βεβαίω όλα τα πολιτικά κόμματα και, και του κρατηδίου, ήμουν και εγώ καλεσμένη και συμφωνήσαμε σχεδόν όλοι ότι τελικά αυτό, αυτή η πρόταση νομοθετική είναι πραγματικά περιττή. Δεν βελτιώνει τίποτα και μάλιστα βλάπτει και την ασφάλεια των επιβατών. Για την προστασία από την ηχορύπανση τώρα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, στη Φραγκφούρτη υπάρχει ένα κίνημα. Στο Αμβούργο επίσης ε, ζω εγώ, στο Αμβούργο είμαι πολύ ικανοποιημένη από την νυχτερινή απαγόρευση που υπάρχει και το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν θα πρέπει να πηγαίνει α, αντίθετα με, τα συμφέροντα των πολιτών και να εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των, α, των ε, αεροπορικών εταιριών. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα για τη, προς την Κομισιόν ε, θέλω να θέσω κι εγώ εκ μέρου ανήσυχων πολιτών πάνω στην πρόταση αυτή για τη μείωση του θορύβου, της χορύπανσης. Υπάρχει φόβος ότι με, την, με τον περιορισμό των πτήσεων τα ε, οικονομικά κριτήρια των ε, ε, αεροπορικών εταιριών θα είναι πολύ πιο σημαντικά από την υγεία τελικά των πολιτών. Η Κομισιόν θα μπορούσε να μας έτσι καθησυχάσει με κάποιο τρόπο. Και άλλο ένα ερώτημα. Υπάρχουν φόβοι σε σχέση με την εξουσιοδότηση που έχει η Κομισιόν την ε, εθνική και περιφερειακή νομοθεσία για τη μείωση των, ε, της συγχωρήβανσης να την ακυρώσει. Η Κομισιόν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ή προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο. Mr. Higgins, two minutes, please. Higgins, δύο λεφτά. Σύντομα σχόλια για την, ε, τις υπηρεσίες εδάφους. καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν. Θέλω να υπάρχει και επιλογή και ανταγωνισμός. Ε, και με καθησυχάζουν αυτά που μας είπε ο κύριος Κάλλας. Ε, και μου αρέσει αυτό που είπε, ότι δεν θέλει να κάνουμε αγώνα για να μειώσουμε τους κανόνες. Ε, αγώνας προς τα κάτω δηλαδή. Αυτό το είπαν και άλλοι, η κυρία Βουίλς και τα λοιπά. Κύριε Διευθυντά, να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η Επιτροπή για τις ε, υπηρεσίες εδάφους. Θα έχει και εκπροσώπους των εταιριών. Συχνά υπάλληλοι του, το προσωπικό εδάφους είναι υπεύθυνοι και για την, την αφαίρεση του πάγου από τις αποσκευές. Δεν θέλουμε μια κατάσταση ε, όπως αυτή που συνέβη τα Χριστούγεννα του 2010. Υπήρχε τέτοιο προσωπικό για να κάνει την αφαίρεση του πάγου και είχαν, υπήρχαν τεράστιες καθυστερήσεις. Όπως είπε και η Κομισιόν, τα, αεροπόρια, τα αεροδρόμια θα πρέπει να συντονίζουν και να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες του προσωπικού εδάφους. Και συμφωνώ με, τα, με όλα όσα είπε σχετικά ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ ο κύριος Φιντάντσα, επίσης δύο λεπτά. Πολύ σύντομα. Για το θέμα των χρονοθυρίδων, συμφωνώ με τις ανησυχίες α, ε, της κ. και άλλων συναδέλφων. Ε, αυτή η νέα διάταξη δεν ξέρω αν μας επιτρέπει να πετύχουμε τους στόχους της α, ε, Κομισιόν, που θέτει η Κομισιόν. Για την δευτερογενή, το δευτερογενές εμπόριο secondary trading. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Μπορεί να χρειαζόμαστε αυτή την ε, πρακτική, αλλά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια από αυτής. Για το θέμα του θορύβου. Η ισορροπημένη προσέγγιση της Κομισιόν είναι ευπρόσδεκτη και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε εδαφικές ιδιαιτερότητες ε, στα πλαίσια της λογικής της ε, επικουρικότητας για την, τις υπηρεσίες εδάφους σε, σε πολλά αεροδρόμια όπου τελευταία έχει επιβληθεί η απελευθέρωση και η εισαγωγή ιδιωτικών εταιριών, έχουμε διαπιστώσει ότι πέφτει το επίπεδο των υπηρεσιών. Θα πρέπει να οπουδήποτε ανοίγει ο ανταγωνισμός, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η σημαντική ευκαιρία που δίνει αυτός ο κανονισμός, ούτως ώστε να αυξήσουμε το επίπεδο των ποιοτικών κανόνων ε, θα πρέπει να επενδύσουμε στις ποιοτικές υπηρεσίες. Ε, όπου, ως λέει και ο κύριος Higgins, δεν πρέπει μόνο απλώς να διαχειριζόμαστε τις αποσκευές. Μιλάμε για πολλές άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει ακόμα και να προβλέψουμε την κατάρτιση του προσωπικού. Ε, πιο πολύ από ό,τι προβλέπει αυτή τη στιγμή το κείμενο της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Για τον οργανισμό, νομίζω ότι δεν ε, καλύπτει επαρκώς τα θέματα της επικουρικότητας. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε κανονισμό. Φοβούμε ότι εάν μία ε, θέτουμε μόνο μέτρα και δεν ε, βάζουμε στόχους, τότε αυτοί που πλήττονται θα είναι σαν να του λέμε ότι οι αρχές τους παίρνουν υπόψη τους ότι υπάρχει θόρυβος, ασχολούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος και ότι τελικά στο τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φταίει που υπάρχει θόρυβος και δεν γίνεται τίποτα για να μειωθεί. Νομίζω ότι η ευθύνη είναι σημαντική και θα πρέπει να την αναλάβουμε. Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένο. Τώρα για τις, ε, τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχουμε καλύτερες και πιο ασφαλείς υπηρεσίες εδάφους. Και κατά την άποψή μου αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο εάν έχουμε καλύτερο προσωπικό, πιο εκπαιδευμένο προσωπικό, με καλύτερο μισθό προσωπικό, ώστε να είναι και καλύτερο γενικά το προσωπικό. Ε, και κυρίως ας πούμε σε μεγάλα αεροδρόμια, σε, αστικούς, ε, σε αστικές ζώνες. Ε, Αυτό που έχουμε θέλουμε να το πετύχουμε και με τον τρόπο που το ακολουθούμε δεν θα το ε, πετύχουμε. Δεν μπορεί κάποιος να εκπαιδεύεται μόνο για δύο μέρες για να προσφέρει υπηρεσίες εδάφους. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά προβληματικό. Οπότε, στο τέλος, θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε τρεις ε, παρόχους με τόσο πολύ περιορισμένα κριτήρια που τελικά δεν θα προσφέρουν τίποτα. Δεν θα προσφέρουν δηλαδή τίποτα που να καλύπτεται από όλα τα κριτήρια ασφάλειας που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ δύο λόγια. Εγώ φοβάμαι για αυτή την κούρσα προς τα κάτω. Το ανέφεραν και ο κύριος Χίγκινς και ο κύριος Φιντάντσα να μην γίνει εξομοίωση με τις χειρότερες προδιαγραφές. Είχαμε όμως αυτή την εμπειρία στο παρελθόν, μία κούρσα προς τα κάτω, προς τα πίσω, όχι μόνο για τις ε, συνθήκες παροχής υπηρεσιών, αλλά και για την ίδια την ποιότητα των υπηρεσιών. Και αποκορύφωμα ήταν αυτό, αυτό το φιάσκο στο Λονδίνο, στο Χιθρό και στις Βρυξέλλες ε, εξαιτίας του υπερβολικού ψύχους. Και το θέμα των υπηρεσιών εδάφους είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να καθησυχάσουμε τα κράτη-μέλη, γιατί στο παρελθόν δεν είχαμε ε, θετικές ε, εξελίξεις. Τώρα για τις χρονοθυρίδες και την δευτερογενή εμπόρια. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτη αυτή η δευτερογενή εμπόρια, το δευτερογενές εμπόριο χρονοθυρίδων. Τώρα για το 85-15 τις αναλογίες έχω κάποιο προβληματισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι το ποσοστό είναι υποδιαπραγμάτευση. Εγώ ε, θα προτιμούσα να εμείνουμε στην ε, Διεθνή Συμφωνία για το 80-20%. Τώρα για το επίπεδο θορύβου και την ηχορύπηση. Εγώ δεν είμαι και κανένα φοβερό υπέρμαχο τη επικουρικότητα, κανονικά τουλάχιστον, φυσιολογικά, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι τοπικέ συμφωνίε, τι τοπικέ συνθήκε για την ηχορύπανση και τα επίπεδα θορύβου. Θα δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις του δικού μας συγκητού για τα επίπεδα θορύβου και θα το συζητήσουμε. Πάντως, το βασικό μου πρόβλημα είναι με τις υπηρεσίες εδάφους και την ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουμε σκανδαλιστεί από την υποβάθμιση αυτών των υπηρεσιών. Και ο χρόνος που περιμένει τις αποσκευές του επιβάτης ε, είναι από τα πιο σοβαρά τώρα θέματα απόψυξης, ε, χρήση αποψυκτικού υλικού για τα αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι ελλείψεις και αδυναμίες των υπηρεσιών εδάφους. Κύριε Μπόλντουιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόσο χρόνο μου διαθέτετε. Δέκα λεπτά κύριε Μπάλντουιν. Ε, γιατί αν τα παρατραβήξετε και πάτε στο τέταρτο θα με φέρετε σε δύσκολη θέση. Καλώς, θα είμαι όσο πιο λακωνικός γίνεται. Για να μην φανώ ότι είμαι άπλιστο στο χρόνο. Βρισκόμαστε, παραλαμβάνω, στην αφετηρία αυτής της διαδικασίας και θα έχουμε πολλές ευκαιρίες. Φάνηκε σημερινή, ε, από τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων ότι επιθυμούμε στενή συνεργασία και με τους ηγητές σας και με την Επιτροπή σας γενικά. Θα ακούσουμε όλες τις πλευρές της βιομηχανίας, τους εργαζόμενους, ε, τους ενδιαφερόμενους, ε, τους επιβάτες. Είχαμε και μία μελέτη επιπτώσεων. Πιστεύω ότι η πρόταση θα είναι ισορροπημένη και σωστή. Φυσικά υπάρχει περιθώριο για αλλαγές και σας διαβεβαιώ ότι είμαστε ανοιχτοί προς τη συζήτηση και τη συνεργασία μαζί σας. Τώρα να συμπληρώσω τις α, ε, απαντήσεις του Επιτρόπου. Καταρχήν, να πω κάποια γενικά και μετά να απαντήσω στις επιμέρους ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τις χρονοθυρίδες, τα σλότς, πολλοί ευρωβουλευτές είπαν ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω μελέτη της κατάστασης. Σας παραπέμπω όμως στην ευρυθέστατη μελέτη ε, της ε, εταιρεία ε, Συμβούλων Steer Davis που πραγματικά ασχολήθηκε εξονυχιστικά με το θέμα. νομίζω ότι ο κύριος Σούτζας, λυπάμαι να προφέρω λάθος το όνομά σας και κάποιος άλλος ζήτησε να σας παράσχουμε όλες τις πηγές μας. Πολύ ευχαρίστω. Αλλά παρακαλώ να σας παραπέμπω στην ε, μελέτη τη Care Agency, πολύ εξονυχιστική μελέτη. Τώρα, σε ό,τι φορά το, την αναλογία για το δευτερογενές εμπόριο των χρονοθυρίδων, το 80-20, 85-15, η μελέτη που σας ανέφερα ασχολείται ενδελεχώ και με το θέμα αυτό. Έχουμε την αίσθηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι αεροπορικέ εταιρείε θα πρέπει εμπράκτο και όχι μόνο με τα λόγια να αποδείξουν ότι χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τι χρονοθυρίδε. Γιατί ε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρω τα σλότ πρώτα. Αυτό το είπε ο Επίτροπο Κάλλα και σίγουρα θα συνεχιστούν ε, οι σφοδρέ συζητήσει για το θέμα αυτό. Για τα επίπεδα θορύβου, η χορύπανση. Ο πρωτορχικό μα στόχο εδώ είναι η διαφάνεια. Και η διαδικασία φυσικά είναι διαφανής θέλουμε. Δεν θέλουμε στόχους ή κατόφλια. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα, τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και για να είμαστε και δίκαιοι, αυτό, γι' αυτό ακούμε και τις περισσότερες μορφές από όλες τις πλευρές. Επίσης προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε την ε, υπάρχουσα νομοθεσία ευθυγραμμίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να καλύψουμε το θέμα της συγχωρήπανσης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαστε απόλυτα συμβατοί με την ισορροπημένη προσέγγιση της ε, Διεθνούς ε, ε, Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Και αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μία προσέγγιση που θα συνάδει με τη διεθνή τάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαδραματίσει μόνο εκ των προτέρων τον ελεκτικό της ρόλο. Θέλουμε να εφαρμοστούν ήδη από την αρχή οι σωστές αποφάσεις, ε, οι σωστές διαδικασίες για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσουμε τα κράτη-μέλη στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Θέλουμε φυσικά να εγκρίνουμε τον κανονισμό, όχι οδηγία, και ο στόχος που προτιμούμε κανονισμό από οδηγία είναι γιατί διαπιστώσαμε κάποιες ασυνέπειες στον τρόπο εφαρμογής των περιορισμών ανά την Ευρώπη. Και μερικές φορές ε, τα επίπεδα θορύβου δεν, συνάδουν με τις ε, προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία. Είμαστε υπέρ της λήψης αποφάσεων, αλλά δεν χρειάζεται να τις λάβει και καλά τις αποφάσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες εδάφους, είναι ένα θέμα που ε, επισημάθηκε από πολλούς. Καταρχήν το ζήτημα της ποιότητας. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρότασή μας όχι ε, μόνο πρόκειται, αλλά η, οφείλει να ευελτιώσει τις προδιαγραφές ποιότητας για τους εξής κύριους λόγους. Ε, δεν έχουμε επαρκή ανταγωνισμό στις υπηρεσίες εδάφους και έχουμε ε, περίτρανες αποδείξεις ότι με τις νέες προτάσεις θα βελτιωθεί και η εμπιστοσύνη των πελατών προς, τους, εταιρείε. Ε, και τα θέματα ευθύνη θα πρέπει να βελτιωθούν, προσαρμογής, μέτρα ασφάλειας όλα αυτά τα μέτρα θα ληφθούν υπόψη, θα προταθούν και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το διαχειριστικό σώμα των μεγάλων αεροδρομίων θα ε, αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ε, θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας ό,τι αφορά τις υπηρεσίες εδάφους. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Μια στιγμή να ολοκληρώσω και θα επανέλθουμε σε λεπτομέρειες. Αυτό είναι ένα από τα προτινόμενα μέτρα που θα βελτιώσει την υψηλή ποιότητα προδιαγραφών. Ακόμη και λόγω κακοκαιρία και διαταραχών τη λειτουργία λόγω κακοκαιρία. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση κατάρτιση, εγώ είμαι υπέρ τη υποχρεωτική κατάρτιση των εργαζομένων. Ένα άλλο μέτρο που στόχο έχει την ε, διασφάλιση υψηλού επίπεδου ποιότητα. Αυτά και τώρα γενικά και έρχομαι προς τα ειδικά σχόλια να ξεκινήσω από αυρότητα από εσά. Και εμά μας απασχολεί και μας φοβίζει αυτή η κούρσα προς τα κάτω. Γι' αυτό και υποβάλαμε τη σχετική πρόταση για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τι εργασιακέ συνθήκες των εργαζομένων, και αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει, για να μην επιδεινωθούν αυτές οι συνθήκες. Και κρατούμε και τα εχέγγυα για του εργαζομένου. Φυσικά θα προσθέσουμε και νέε εγγυήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή ο τρόπος που διαμορφώνεται η νομολογία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να μην απαιτούν από τους νέους παρόχους που ε, απασχολούν το ίδιο προσωπικό με τους προκατόχους τους να, να μην είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, να μην είναι υποχρεωμένοι να απασχολούν δηλαδή τους προηγούμενους ε, εργαζομένους. Εμείς θέλουμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να απαιτούν ε, από τους παρόχους, να κρατούν τους παλιούς εργαζομένους. Ε, νομίζω ότι έτσι έχουμε μια ασφαλιστική δικλίδα για αυτούς που φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους σε περίπτωση που αλλάξει ο πάροχος υπηρεσιών. Και κάθε πάροχος ε, θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις ε, εθνικές διατάξεις κοινωνικής πρόνοιας και τις κοινωνικές και εργασιακές διατάξεις και υπάρχει το θέμα της πιθανότητας υποχρεωτικής κατάρτισης των εργαζομένων και τα ελάχιστη, οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την απασχόληση. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε καλύτερα καταρτισμένο προσωπικό και πιο ασφαλείς θέσεις εργασίας. Τώρα, η κυρία Αγιάλα, λυπάμαι στο μεταξύ, έφυγε, ρώτησε γιατί δεν προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τις υποδομές μας. Αυτό το θέμα το καλύπτουμε σε μια ειδική ανακοίνωση σύντομη απάντηση είναι ότι θέματα υποδομών είναι ευθύνη των κρατών μελών. Πολλοί μπορεί να διαφωνούν για αυτή την αρμοδιότητα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τα κράτη-μέλη επιμένουν να έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για, το, για τις αποφάσεις που θα κατασκευάσουν ένα αυτοκινητόδρομο, θα κατασκευάσουν, αν θα χτίσουν νέο αεροδρόμιο. Αλλά μπορούμε να έχουμε κοινά, κοινές προδιαγραφές ε, για να καταμετρήσουμε το δυναμικό των αεροδρομίων. Πάντως προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη εικόνα για την κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κυρία Γιάλα ρώτησε πώς ο διαχειριστικός φορέας του αεροδρομίου θα εργαστεί σε ό,τι φορά τις υπηρεσίες εδάφους. Σας παραπέμπω στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του πακέτου μας και πολύ ευχαρίστω να επανέλθουμε στη συζήτηση. Ο Νομίζω ότι κάντε μια ερώτηση για τι χρωμοθυρίδε, στην οποία έχω ήδη απαντήσει με τα όσα έχω πει. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ναι, ε, του ε, μικρού αερολιμένε. Ε, Βεβαίω μα ενδιαφέρει αυτό και θα το, θα το λάβουμε υπόψη όταν συζητάμε για τα περιφερειακά δρόμια. Δεν κοιτάμε μόνο του μεγάλου παίκτε. Ο κύριο Κράμερ έκανε διάφορε ερωτήσει για την αεροπορική εταιρεία. Η η αεροπορική εταιρεία μας λέει ότι αυτή πληρώνει για τις ε, υποδομές της. Έτσι πιστεύουν. Και στους άλλους τομείς των μεταφορών, ε, σωστό είναι ότι οι εταιρείες πληρώνουν περισσότερα. Για τα ελάχιστα πρότυπα του θορύβου, ε, απάντησα ήδη. Δεν μπορούμε εμείς η Κομισιόν ή οποιοδήποτε ευρωπαϊκός εδώ πέρα, ευρωπαϊκό όργανο, να επιβάλλει κάποιους κανόνες. Απλώς προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την όλη διαδικασία να πλαισιώσουμε την όλη διαδικασία. Κύριε Κόχ, ε, ερωτήσεις κάνετε για, τον, για την χορύπανση και ανησυχείτε γιατί ε, τα θέματα των χρημάτων, τα οικονομικά, εν και τις παροχές υπηρεσιών θα γίνουν πιο σημαντικά από την υγεία. Ε, εμείς δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάποιες διαδικασίες. Ε, οι, τοπικοί, οι τοπικές αρχές είναι αρμόδιες. δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα εμείς. Επίσης, δεν μπορούμε εμείς ε, να αποφασίσουμε ότι οι εθνικοί κανόνες είναι άκυροι. Ε, η Κομισιόν δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη ε, στις αποφάσεις τους. Κύριε Χίγγινς, μιλήσατε για τη σύνθεση της Επιτροπής Χριστών του Αεροδρομίου. Το άρθρο 4.1 μιλάει για αυτές τις διατάξεις. Μπορώ να το ξανασυζητήσω μαζί σας. Κύριε Γκάλερ. Νομίζω ότι κάλυψα τα ερωτήματα που θέσατε. Αυτά με βάση το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου ε, προσπάθησα να απαντήσω όσο μπορούσα πιο γρήγορα ε, στις άρθμες αυτές σημαντικές ερωτήσεις. Ε, απλώς είναι μια πρώτη συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί μαζί σας και με, άλλα, και με άλλους. Η κυρία Μάισνερ. Η πιο σημαντική ερώτηση δεν απαντήθηκε. Γιατί αναγκαστήκατε να αλλάξετε και να κάνετε κανονισμό αντί για οδηγία. Γιατί ο κανονισμό, όπω ξέρετε, είναι λιγότερο ευέλικτο από την οδηγία. Νομίζω ότι αναφέρθηκε ήδη. ήδη. Θέλετε να το επαναλάβετε, σα παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Μάισνερ. Ίσως το είπα πολύ γρήγορα και πολύ λακωνικά. Πάντως, να επαναλάβω ότι είχαμε διάφορε ανησυχίε για τον θόρυβο Φερρυπίν ότι οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο, με συνεπή τρόπο. Προσπαθούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ίδια εφαρμογή. Θέλουμε ας πούμε οι, οι συνθήκες ας πούμε, ασφάλειας να εφαρμόζονται όταν δεν θέλουμε σε περίπτωση δεν θέλουμε με τον κανονισμό να πούμε ότι αυτό είναι το μοντέλο και το επιβάλλουμε παντού. Απλώς πιστεύουμε ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις καλύτερα μέσω του κανονισμού. Αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπε και ο ομιλητής, είναι η αρχή της διαδικασίας. Θα γίνει μια πολύ μακρά συζήτηση εδώ με τις ομάδες. Σας ευχαριστώ και σας υπενθυμίζω. ότι εξασφαλίσαμε την παρουσία του Επιτρόπου λόγω της καταστροφής με το υπεροκειάνιο, με το κροσγερόπλιο. Η Μπάρα, μία από τις γραμματείς μας, ε, θέλω να σας ότι φεύγει από την Επιτροπή ε, Μεταφορών. Από το 2006 εδώ η Μπάρμπαρα ε, είχε δουλέψει πριν με την Κομισιό, στα, στους κόλπους της Κομισιόν. Άρα δούλεψε και με τους καλούς και με τους κακούς. Και τώρα μπαίνει στο γραφείο του Προέδρου Σούλτς. Μπάρμπαρα, σε ευχαριστούμε για όλη τη βοήθεια. Η Μπάρμπαρα είναι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα παρασκήνια. Δεν φαίνεται ότι κάνει τη δουλειά. Αλλά αυτή οργανώνει τις ε, συνεδριάσεις, ε, κλείνει τις αίθουσες ε, συνεδριάσεων, κάνει το πρόγραμμα. Η Μπάρμπαρα τα κάνει όλα αυτά. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτά τα, τα πρώτα δυόμιση χρόνια της κοινοβουλευτικής θητείας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, Μπάρμπαρα, σου εύχομαι καλή τύχη ε, στη συνεργασία σου με τον πρόεδρο Σούλτς. Και τώρα ξέρουμε το, το μέσο που έχουμε στο γραφείο του Προέδρου, θα το χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Uh, Πάμε στις συνεδρίες των ε, συντονιστών. Σε δύο λεπτά.